Okay. Liebe good morning. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μετά τις διακοπές βλέπω μόνο χαρούμενα πρόσωπα, άνθρωπους ξεκουρασμένους. Ναι, δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει το μικρόφωνο του πρόεδρου. Δουλεύει. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους. Χαίρομαι που ξεκουραστήκατε. Έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα. Να κάνω μία παρατήρηση οργανωτική. Σας παρακαλώ σήμερα να χρησιμοποιεί το μικρόφωνο στα αριστερά, μου είπε ο τεχνικός. Δεν το κατάλαβα, μου είπε, εν πάση περιπτώσει, το αριστερό μικρόφωνο χρησιμοποιείτε. Δεν ξέρω γιατί, έτσι μου είπαν τεχνικοί, κάτι θα ξέρουν. Ε, συνήθως έχω πρόβλημα, εγώ ξέρετε, με τα αριστερά, τα μικρόφωνα ή όχι, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεύτερη παρατήρηση. Τα σημεία 9 και 10 έχουν αλλάξει. Στα σημεία 11 και 12, δηλαδή με τους Βέλγους Υπουργούς ε, είπαμε να ξεκινήσει η συζήτηση 11 και 30 οπότε θα έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας ε, λυπούμε, αλλά αλλιώ δεν γινόταν τίποτα. Και βλέπετε πως είναι τεράστια η ημερήσια διάταξη, οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οπότε παρακαλώ να με βοηθήσετε για να τηρηθεί και ο χρόνος. Το τρίτο για τις ανακοινώσεις ε, του Προέδρου αφορά το θέμα προφορικές ερωτήσεις για την κλιματική διάσκεψη. Ε, επίθυνα μια επιστολή τέλος Ιουνίου στον ε, συνάδελφο της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος δεν, για να το κάνουμε μαζί δεν έχω λάβει απάντηση αλλά ξέρω πως θέλει να κατατεθεί προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια και πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Δεν ξέρω γιατί είναι μόνο υπόθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και εγώ προτείνω να το δούμε αυτό στο σημείο 13 και να καταθέσουμε και εμείς Αποκινούμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος το προφορικό ερώτημα για να είναι κενό. Οπότε θα σας παρακαλέσω να το ξαναδούμε στο σημείο 13 και τέλος έχουμε και το ερώτημα προς την κυρία Κρούς για τα δίκτυα επόμενης γενιάς. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση οπότε νομίζω πως η επιστολή μπορεί να αποσταλεί ως έχει. Παρακαλώ, έχετε πρώτο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας υπόψη το ότι δεν θα συνεδριάσουν οι συντονιστές παρά μόνο την επόμενη φορά. Και θέλω να σας επισημάνω κάτι το οποίο μου υπέδειξαν χτες σε μια συνεδρίαση με εκπροσώπους του κλάδου της βιομηχανίας συγκεκριμένα από την αεροδιαστημική για το REACH και για ένα θέμα για το οποίο εν μέρει ήταν ε, σαρμόδια η Επιτροπή ε, και είχαμε συνεργαστεί με την περιβάλλοντα επίση, Το πρόβλημα ήταν η καταχώρηση κάποιων χημικών ουσιών, η προθεσμία του Δεκεμβρίου και η φόβη τη βιομηχανία ότι υπάρχουν κάποιες χημικές ουσίες που σήμερα είναι αναντικατάστατε και ότι πρόκειται να αποσυρθούν από την αγορά. Δεν θέλω τώρα να προκαλέσω συζήτηση. Σήμερα, Πρόεδρε, όμως, αυτό ενδεχομένω είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τη βιομηχανία. Γι' αυτό σα προτείνω να καλέσουμε την Επιτροπή να έρθει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή μα και να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων γι' αυτό το θέμα και να μα ενημερώσουν σε σχέση με το πώ πάνε και τα πράγματα γιατί δεν θέλουμε να αναγκαστούν ε, ένα σωρό εργαζόμενοι να πάνε εκτό Ευρώπη να δουλέψουν και αυτό διότι υπάρχει παρερμηνία ή τέλο πάντων δυσχερή ερμηνεία ενός νομοθετήματος. Παρακαλώ λάβετε το αυτό υπόψη και προσπαθήστε να καλέσετε σε λίγες εβδομάδες την Επιτροπή για να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα αυτό. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστώ. Το έχουμε συζητήσει ήδη μία φορά αυτό το θέμα. Είχαμε πληροφορηθεί πως είμαστε σε καλό δρόμο. Εάν συμφωνείτε όμως τώρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε γιατί δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Εάν λοιπόν δεν έχει κάποια, κάποια αντίρρηση κάνουμε δεκτή την πρόταση Τσίτσεστερ και θα προσκαλέσουμε τους κυρίους αυτούς σε μια επόμενη συνεδρίαση. Αν συμφωνεί και η γραμματεία, ωραία. Λοιπόν, α, ε, τώρα δεν, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση, λίγο γρήγορα άμα είναι, σε παρακαλώ. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό που μας είπε ο Τσάλης πριν από λίγο, όμως όταν έρθει η Επιτροπή, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια γενική συζήτηση σε σχέση με το πώς τα πράγματα γενικότερα με το Ρίτς και όχι μόνο με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Also, Εντάξει λοιπόν, ξεκάθαρο. Σημεία 3. Α, Παουλ Ρούμπιχ, ναι, ε, τώρα ξεκίνησαν όλοι. Ναι, για αυτό το οποίο ανέφερες για τα δίκτυο της επόμενης γενιάς για την επιστολή Κρούς, πρέπει να γράψουμε πως και οι στόχοι πρέπει να είναι πως δεν θα έχουμε πλέον καθόλου τέλη περιαγωγής αλλά να ισχύσει επιτέλους η εσωτερική αγορά. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό. Ε, κοιτάξτε, αυτό θα το αλλάξω αν συμφωνούν όλοι, αλλά δεν είναι όλοι εδώ. Οπότε θα το στείλω με email στους συντονιστές ε, και θα δούμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Εντάξει, το άκουσα αυτό που είπατε, θα στείλω email και τα Εάν έχει ένα αντίρρηση δεν θα μπει βεβαίω λοιπόν. Οντί. Εντάξει. Ναι, ναι, τακτοποιήθηκε. Ωραία. Ευχαριστώ. Σημείο 3. Μιλάμε για έγκριση πρακτικών της ε, συνεδρίας της 1ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου και 23 και 24 Ιουνίου. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 4, διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων. Να σας πω, έχουμε 15 λεπτά για αυτό το θέμα και θα είμαι πολύ αυστηρός σήμερα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το λόγο έχει ο συντάκτης γνωμοδότησης ο κύριος Τζάιλς Τσίτσεστερ. Έχετε τον λόγο. Uh, thank you, Chairman. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μισό λεφτάκι για να βρω τα χαρτιά. Το θέμα αυτής της αξιολόγηση και διασφάλιση εκτιμήσεων ε, είναι ένα θέμα το οποίο σε μένα αλλά και τη συνάδελφα Αγγέλη Γανίμπλερ για μια άλλη επιτροπή. Εγώ έχω συντάξει ένα σχέδιο κειμένου που δεν είναι ουσιαστικά σχέδιο γιατί ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και μετά θα το ολοκληρώσουμε και τότε θα το στείλουμε για μετάφραση πάντως. Είναι έγγραφο για συζήτηση. Το θέμα είναι απλό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εκτίμηση επιπτώσεων στα νομοθετήματα. Ναι, βέβαια. Και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να γίνει. Το δε επόμενο θέμα είναι πιο σοβαρό. Ποιος θα πρέπει να κάνει αυτές τις αξιολογίες επιπτώσεων γιατί μέχρι τώρα τις έκανε η Κομισιόν. Και η Κομισιόν έχει ένα σωρό ικανούς υπαλλήλους. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι έχουν συντάξει και την πρόταση. Ε, οπότε έτσι υποβαθμίζεται η μελέτη των επιπτώσεων, εάν την κάνουν οι ίδιοι. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι η ουσία αυτού του κειμένου μου είναι να μπορέσω να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ανεξάρτητη τέτοια μελέτη. Αυτό λοιπόν θέλουμε να προτείνουμε και να εφαρμοστεί και γι' αυτό καλό τους συναδέλφους να διαβάσουν αυτό το κείμενο, είτε το λέμε σχεδόν κειμένο ότι όχι και έτσι καλώς έχουμε μια εβδομάδα, μέχρι την εβδομάδα τέλος πάντων για να το στείλουμε στην μετάφραση Οπότε, αν είναι δυνατόν, να μπορέσω να καλύψω ό,τι θα μου προτείνουν. Και να λάβω υπόψη το ότι υπάρχουν ένα σωρό προτάσεις που θα πρέπει αργότερα να τις ε, προωθήσουμε και έχουμε και ενδεχομένω κάποιες τροπολογίες που και έτσι μπορούμε τελικά να ξεπεράσουμε τον περιορισμό για την έκταση του εγγράφου ο οποίο υπάρχει. Αυτό είναι το βασικό θέμα. το πώ θα είναι επομένω ανεξάρτητα σε αυτέ οι μελέτες επιπτώσεων και πώ, η Κομισιόν μα εξηγήσει ε, γιατί πρέπει να γίνει, να μην γίνει, να υπάρχει διαφάνεια σχέση με αυτό και ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κατά την νομοθετική διαδικασία ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη ενημερώνοντας αυτές τις μελέτες το τι λέει το Συμβούλιο ή τι λέει τα διάρκεια διαδικασία στο Κοινοβούλιο. Και ζητώ να εγκρίνετε την πρότασή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος τον λόγο. Κυρία Μαδουρέλα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σαν σκιώδης εισηγήτρια παρεμβαίνω από την ομάδα μου για το θέμα αυτό. Να σας πω ξεκινώντας ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη τεράστια προσπάθεια και την πρόοδο της Επιτροπής τα πέντε αυτά τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα πλαίσια, δηλαδή σε αυτό που λέμε better law making, ε, καλύτερη νομοθεσία. Έτσι και με περισσότερο διάφωνο, αποτελεσματικό, σαφή, συγκεκριμένο, ισορροπημένο τρόπο. Να σας πω επίσης ότι σήμερα η ομάδα μου αυτή την εκτίμηση του κ. στο εγγραφό του εδώ για τη σημασία αυτών των εξελίξεων και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την ομοθετική μας εργασία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτές τις μελέτες που είναι απαραίτητες για να πετύχουμε και το Small Business Act. Εδώ να σας πω ότι παραμένει ένα αρκετά σημαντικό περιθώριο λιγμών για να βελτιώσουμε στο σύνολό του αυτές τις καταστάσεις και αυτές τις μελέτες και για να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά εφαρμόζονται συγκεκριμένα και αποτελεσματικά. Και σαν ε, Γενική Αρχή υποστηρίζουμε ότι με τη δική μας την οργάνωση, με την Επιτροπή Εκτίμησης των Επιπτώσεων, ε, ε, εδώ αναφέρει κάτι το πιο ριζοσπαστικό ο κύριος Τσίσεστερ και που μας παρουσίασε τώρα. Ε, συμπίπτουν οι απόψεις μας ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε βέβαια την σημερινή διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή και θα πρέπει να δούμε αυτές τις πτυχές όπως την διαφάνεια και τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας πάντα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα όπως αυτά που θα πω στη συνέχεια να δημοσιευθούν και να υπάρξει μια διαβούλευση για τις μελέτες επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της ε, ε, εξέτασης αυτής νομοθετικής ε, της διαδικασίας και επίσης με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπάρξει μια επαφή για τους ίδιους λόγους επίσης να υπάρξει μακρύτερη περίοδος τουλάχιστον δύο εβδομάδες για τη διαβούλευση και ακόμα κάτι τελευταίο, κάτι το απαραίτητο που θα ήθελα να τονίσω είναι οι πτυχές περί περιβάλλοντος και κοινωνικές πτυχές να ενσωματωθούν στην ε, μελέτη επιπτώσεων και διαθέτουμε πείρα και βλέπουμε ότι γιατί αυτές οι εκτιμήσεις επιπτώσεων δεν θα πρέπει να περιστούν μόνο στις οικονομικές επιπτώσεις. Ε, όπως είπε ο κύριο Τσίστεστερ κύριε Πρόεδρε, η συνάδελφος Άντζελα Μνίμπλερ, εξέχον μέλος, ε, είναι με την τύχη που είναι εισηγήτρια και διάβασα το έγγραφο εργασίας της, όπως επίσης ε, και τα θέματα που θέτει και που είναι αυτά που πρέπει να εξετάσουμε, θα πρέπει να υποφεληθούμε και από κοινού επεξεργαστούμε το θέμα αυτό. Όπως και η συγγήτρια ε, ε, το λέει, θα συνεργαστούμε και εμείς για τις καλύτερες προτάσεις ε, για αυτές τις μελέτες επιπτώσεων και πώς όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νίμπλερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και τον κύριο Τσίτσεστερ που έχει κάνει εδώ πέρα ένα πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης όπως και την κυρία Ριέρα Μαδουρέλ για τις πολλές προτάσεις βελτίωσης για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων αλλά και για το τι μπορούμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο. Μπορώ να υποστηρίξω πάρα πολλά πράγματα και νομίζω πως βοηθούν πάρα πολύ αυτές οι ιδέες. Σημαντικό είναι να έχουμε κατά νου πως οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καλύτερης νομοθεσίας. Έχουμε πολλές εμπειρίες, λοιπόν. Σωστά διαπιστώνουμε πως εντός της ε, Κομισιόν οι εκτιμήσεις επιπτώσεων έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Προσπαθούν να τις κάνουν ανεξάρτητες, αλλά όπως βλέπω και όπως λένε και οι συνάδελφοι εδώ πέρα χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, βελτίωση, μια πιο ανοιχτή διαδικασία για να διασφαλίσουμε και να εξηγήσουμε ε, εάν δεν υπάρχει κάποια τέτοια αξιολόγηση γιατί έγινε αυτό. Και ο κύριος ε, Τσίτσεστερ νομίζω είπε τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω πως ε, το κάνουν ήδη κάποιες επιτροπές. Δηλαδή όταν έχουμε σοβαρές προτάσεις αλλαγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν πρακτικές επιπτώσεις και σήμερα ούτως ή άλλως μπορούμε ανεξάρτητα να παραγγείλουμε μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων. Το θυμάμαι και με την κυρία Ριέρα Μαδουρέλ που είμαστε μέλη στην Επιτροπή Γυναικών που είχαμε αυτή την οδηγία την προστασία της μητρότητας πριν από την ολοκλήρωση πρώτης ανάγνωσης ζητήσαμε εκτίμηση επιπτώσεων λόγω των αλλαγών που προτείνονταν. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε το τι άλλο μπορεί να γίνει. Και ο κύριος ε, Τσίτσεστερ νομίζω είπε πως θα πρέπει να μπει και το ελεγκτικό συνέδριο στην όλη διαδικασία και αυτό ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συζήτηση και αναμένω βεβαίω και την πρόταση στην οποία θα δείξει η νομοδότηση Τσίτσεστερ και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα μεταφέρω οπωσδήποτε τα επιχειρήματα της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μας. Ε, ε, Αυτή η συζήτηση για καλύτερη νομοθεσία φαίνεται να είναι καθαρά τεχνοκρατικό θέμα. Σας υπενθυμίζω όμως ότι είναι πολιτικό και πολύ πολιτικό μάλιστα. Η πρώτη επιτροπή Μπαρόσου και πάρα πολλοί επιχειρηματίε. επαναλαμβάνουν ότι αν δεν έχουμε καλύτερη νομοθεσία, να μην έχουμε καθόλου νομοθεσία και σα λέω ότι τι γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με τι επιχειρήσει στην Κομισιόν. Ο κ. Στόμπερ λέει ότι πρόκειται για ένα βάρο τη βιομηχανία, τη επιχειρήσει και θα πρέπει να έχουμε όσο γίνεται λιγότερη νομοθεσία. Όσο γίνεται λιγότερη. Επομένω, ε, μπορείτε έτσι να πάρετε μια πρόγευση για το περί πρόκειται. Οπότε, θα πρέπει όλους όσους διαμορφώνουν την πολιτική να τους ε, προειδοποιήσω ότι μετά από 10-15 χρόνια ε, που έχουμε αυτή την αόρατη χείρα η οποία ρυθμίζει τα του τραπεζικού κλάδου Μα διαπιστώσει κανεί εύκολα όταν δει πώς έχει εξελιχθεί το θέμα τα τελευταία διετία, τριετία. Όλοι αυτοί που θέλουν βολονταρισμό εκεί και τώρα διαμορφώνουν το πλαίσιο των ρυθμίσεων στον τραπεζικό κλάδο. Όλα αυτά επομένω μας οδηγούν στο να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι στο σημερινό κόσμο χρειάζονται κάποιοι να διαμορφώνουν την πολιτική με τους σωστούς κανόνες. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι η κοινωτική νομοθεσία αντικαθιστά όλους εκείνους τους νόμους των 27 κρατών μελών. Άρα, εξορισμού πρόκειται για μείωση του διοικητικού βάρους, γιατί έτσι κάνει ευκολότερη τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και αυτή που δεν πράγμα την πολιτική να είναι ελεύθερη αλλά λάβουν υπόψη ε, κάθε τροπολογία μας γιατί φυσικά και δεν είναι ακριβής επιστήμη η χάραξη πολιτικής και ξέρουμε ακριβώς και αυτό είναι ακριβώς το καλό το ότι εδώ έχουμε πολλές διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι θέλουν η αυτοκινητοβιομηχανία να έχει πιο αυστηρούς κανόνες γιατί ακριβώς έχουμε το ενεργειακό, έχουμε έναν πλανήτη όπου αν έχουμε ξαφνικά δύο-τρία δις ε, αν θέλουν τα πάρουμε και ε, δεν θα τους αντέξει ο πλανήτη. Άρα έχουμε αυτού που χάσουν την πολιτική οι οποίοι τι θέλουν. Θέλουν να συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις τεράστιες λιμουζίνες. Επομένως δεν καταλαβαίνω πώς κάποιο ε, στην διοίκηση του Κοινοβουλίου θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Είναι ψευδέστηση το πώς θα χτενιστούν οι τροπολογίες. Είχαμε 1500 τροπολογίες όταν εγώ έκανα εκείνη την έκθεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένω, θα πρέπει να χτενιστούν όλες οι τροπολογίες. Άρα φυσικά και θέλουμε στοχευμένες ερωτήσεις, θέλουμε κάποιες συμβουλές, θέλουμε σε κάποια συγκεκριμένα θέματα συμβουλές, αλλά να μην μας δέσει χέρια και πόδια κάποιος Σύμβουλο σε κάποιο απομονωμένο γραφείο θεωρώντας ότι είναι σοφότερος, εξυπνότερος από εμάς. Και αυτή τώρα εξωτερική ειδική είναι κάτι το ενδιαφέρον να, να δούμε ποιος τους θέλει Ποιο θέλει να του βάλει δίπλα στον κάθε υπάλληλο οποιασδήποτε επιτροπή που θέλει να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Έχουμε εδώ πέρα το ΑΣΕΑ, είναι μια ουδέτερη ε, οργάνωση γενικού ε, με γενικά ενδιαφέροντα, γενικέ αρμοδιότητε και ζητά εξωτερικούς συμβούλου, οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν και να αντικαταστήσουν αυτού οι οποίοι κρίνουν και δημορφώνουν την πολιτική στην Ευρώπη. Και γι' αυτό σας προειδοποιώ, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τελευταία παρατηρήση τώρα. Πάρα πολύ δεξιοί που διαμορφώνουν τις πολιτικές, πάντοτε, πάντοτε, λαμβάνει υπόψη τι γίνεται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Για να κοιτάξτε όμως και σε αυτή την περίπτωση, και εδώ θα διαπιστώσετε ότι στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε προβληματίζονται πάρα πολύ όσον αφορά την καλύτερη νομοθεσία και το Κογκρέσο κατέληξε στο ότι είναι αδύνατον να ελεγχθεί η κάθε τροπολογία που υποβάλλεται για κάθε νομοθέτημα και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουν είναι το να παρακολουθούν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτή είναι η προσθεμενή αξία. Πολλέ φορέ έχουμε πολύ καλή κοινωνική νομοθεσία, αλλά δεν μεταφέρεται στο ιστορικό δίκαιο σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πώ εφαρμόζεται η κοινωνική νομοθεσία. Αυτό θα είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία. Οπότε τελείωσε και αυτή η συζήτηση. Α, ναι. Ε, ποιος, δεν ξέρω. Και ο, ο Σοντή, ορίστε. Δεν αντέχω, πρέπει να παρέμβω μετά από αυτή τη σκιαγράφηση με αυτόν τον τρόπο. Όταν θέλει κανείς να καταστραφεί, έχουμε την πρώτη μέθοδο να παίξει μετά, ε, είτε να ασχοληθεί με γυναίκες και αυτή είναι πιο ευχάριστη και μετά να ακούσει τους εμπειρογνώμονες. Ε, τρεις μέθοδοι για να αυτοκαταστραφεί κανείς. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δούμε ποτέ η... Ε, τα άτομα αυτά δεν έμειναν ανεξάρτητα. Δεν είμαστε όπως οι Αμερικανοί με 30-40 συμβόλους έχουμε, λόμπι γύρω έχουμε όλα αυτά. Εγώ βέβαια χαίρομαι για την εργασία του συνάδελφου ε, Τσίσεστερ ενώ το Στόιμπερκ εντάξει βλέπω διάφορα κενά, διάφορες ελλείψεις του σε πολλά θέματα που ε, συζητήσαμε σε άλλους χώρους αλλά θέλησα να κάνω αυτή, πρέπει σε αυτή την καρικατούρα πάνω που άκουσα, που είδα. Ευχαριστώ. Και τελειώνει εδώ η συζήτηση. Όπως πάντα στη ζωή οι απόψεις διαφέρουν. Άλλοι θένε περισσότερη ρύθμιση, άλλοι λιγότερη. Ε, μπορούμε να συζητάμε για πάντα. Λοιπόν, ο Τζάιλ ο ο έχει το δικαίωμα να επανέλθει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι η Κομισιόν σε αυτό το σημείο. Ε, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ υπερβολικά ίσως γιατί αυτό το έγγραφο το οποίο έχετε λάβει δεν είναι το οριστικό. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι για την ανταπόκριση και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και την υποστήριξή τους. Τη Λουίζα Μαντουρέλ δεν κατάλαβα αν είναι μαζί μου ή εναντίον μου. Θα τα δούμε πάντως σε λεπτομέρειες του τα θέματα και πάντως νομίζω ότι πάρα πολύ χρήσιμο να βελτιώσουμε το κείμενο. Επίσης θα πρέπει να συγχαρώ τον Κλοντ Τούρμες γιατί πάρα πολύ κομψά ε, ε, έστειλε τη σύντηση προς την άλλη κατεύθυνση προς την προβληματική του φθινοπόρου, την αντιπαράθεση δεξιάς αριστεράς. Αυτό έχει ενδιαφέρον, έχει πλάκα και τον ευχαριστώ. Αλλά νομίζω ότι ε, είναι λίγο σκληρός, λίγο αυστηρό με τον κύριο Λάγκεν γιατί περισσότερο μας νομίζω συμφωνούμε ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι η πρόθυμη θέσπιση καλύτερης νομοθεσίας. Περιστάσεις αλλάζουν και θα πρέπει να δούμε πώς έχουμε κοινέ απόψεις πρασίνων και άλλων για κάποια σημαντικά θέματα. Τώρα, σε συνέχεια κάποιου συγκεκριμένου θέματος, δύο-δύο, σε δύο σημεία όπω αναφέρθηκε ο Κλοντ, να πω τα εξή. Πρώτα-πρώτα, περιγράφει την κοινοτική νομοθεσία ότι αντικαθιστά πάρα πολύ ε, πάρα πολλά εθνικά νομοθετήματα. Μόνο σημαίνει λιγότερη νομοθεσία. Όμω ε, θέλω να σου πω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το αντίθετο. Ότι η κοινωτική νομοθεσία προκαλεί βουνά νόμων εθνικών Βρετανικών γιατί παίρνουν οι βουλευτές κάποια οδηγία 12-20 σελίδων και ακριβώς επειδή ε, θέλουν όλα να τηρηθούν και τελευταία κεραία του κοινωνικού κειμένου φτιάχνουν ένα νομοθέτημα εκατοντάδων σελίδων Επομένω, πάρα πολύ αξιέπαινο το είπε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικά. Κάτι άλλο, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε, ε, ότι είσαι δηλαδή κατά των εξωτερικών συμβούλων. Όχι. Δεν χρειάζεται να είναι εμπειρογνώμονε. Απλώ εμεί θέλουμε μια ξεχωριστή ε, μελέτη αναθεώρηση των κειμένων. Και όσον αφορά το ότι είσαι κατά αυτών των ανεξαρτήτων ε, συμβούλων, ανέφερε και την αυτοκινητοβιομηχανία και νομίζω ότι εσείς πρώτοι, οι πράσινοι, χρησιμοποιείτε συνέχεια ειδικού. Παρά ότι είστε οι ίδιοι ειδικοί για τα θέματά σας. Ε, λοιπόν, για να τα προωθήσετε, καλείτε εξωτερικού εμπειρογνώμονε. Μπράβο, θα πρέπει πάντα να έχουμε τις διαφορετικές ε, ε εναλλακτικέ για να δούμε πώς θα προωθήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μιλάμε για απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίου για την έρευνα. Έχουμε όμως και άλλο ένα σημείο πριν την ψηφοφορία, οπότε παρακαλώ να προσέξουμε να τελειώσουμε και τα δύο αυτά θέματα. Λοιπόν, η κυρία Καρβάλιο είναι υπεύθυνη. Έχουμε επίσης και επισκέπτες από την Ισπανία, του οποίους καλώς ορίζω. Λοιπόν, κύριε Καρβάλιο, έχετε τον λόγο. Α, από την Πορτογαλία. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, τρομερό λάθος, συγγνώμη. Thank you. Thank you, President. Uh, good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank uh, all my colleagues να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους για τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει στην έκθεσή μου και ευχαριστώ για το πόσο βοήθησαν την ουσία της έκθεσής μου και θέλω σήμερα να σας πω κάποιες γενικές παρατηρίες για αυτές τις τροπολογίες στη συνέχεια δε να σας πω γιατί θεωρώ ότι πρέπει να γίνει με αυτές τρεις κατηγορίες των προτάσεων. Τέλος, να δούμε ε, πώς βουνάρουμε κάποιες αντιφάσεις που έχουν οι τροπολογίες. Τέσσερα σημεία πρώτα-πρώτα, οι περισσότερες από τις τροπολογίες προσθέτουν νέες ιδέες σε αυτή την έκθεση. Πουθενά δεν επικοινωνούνται οι βασικές προτάσεις της έκθεσης. Έτσι, θα συμπληρώσουμε το σχέδιο με κάποιες προτάσεις που δεν υπάρχουν στο πρώτο σχέδιο Δεν είχαμε το, το, το, το χώρο για να τα καλύψουμε, αλλά δεν υπάρχουν επομένω ε, αντιθέσει μεταξύ των βασικών πολιτικών ομάδων και μπορούμε να έχουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες τροπολογιών εδώ. Πρώτα-πρώτα κάποιες οι οποίε έχουν κάποιες καινούργιες προτάσεις. Ε, είμαι υπέρ. Δεύτερον, έχουμε κάποιες που έχουν να κάνουν με κάποιες προτάσεις που ήδη υπάρχουν στην έκθεση και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τις καλύψω όλες αυτές με συμβαστικές τροπολογίες. Είναι και κάποιες όμως που βρίσκονται εκτός θέματος. Αυτές είναι ακόμα ένα βήμα σε αυτή την πορεία για την ολοκλήρωση, την έγκριση του προγράμματος πλαισίου. Και τώρα, τρίτο σημείο, τα επίμαχα θέματα. Θα πρέπει τα εξής τέσσερα θέματα να λάβουμε υπόψη. Πρώτα-πρώτα, προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων. Εδώ έχουμε τροπολογίες που αντιφάσκουν, ορισμένες τροπολογίες είναι υπέρ αυτής της μεθόδου και κάποιοι συνάδελφοι θέλουν ε, περισσότερη ανεξάρτητη έρευνα από την βάση προς την κορυφή και να υπάρχει μια προσέγγιση που να αντιμετωπίζει τους κινδύνους ε, και με μηδέ εμπιστοσύνη βασίζεται σε επιστημονικές απόψεις. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια διάκριση μεταξύ πανεπιστημίων, ΜΜΕ και βιομηχανίας. Όμως κάποιοι συνάδελφοι προτιμούν μια ενιαία αντιμετώπιση από όλους για διαχείριση, διάχυση αποτελεσμάτων κλπ. Εδώ μπορούμε να βάλουμε μια ε, τροπολογία συμβαστική που να λέει για το πώς θα έχουμε μια μείωση των, ε, ε, των κριτηρίων αλλά όχι όμως μόνο ένα για όλες τις δραστηριότητες. Τώρα όσον αφορά κάποια φάπαξ ποσά έχουμε κάποιες κάποιες τροπολογίες που θέλουν υπάρχουν ε, ποσά ε, τα οποία να είναι φάπαξ εννοώ ενιαία αλλά κάποια άλλοι όχι οπότε ε, εγώ νομίζω θα πρέπει κάθε θεσμικό όργανο να μπορεί να διαλέξει ποια μέθοδο προτιμάει επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες τροπολογίες που σχετίζονται με τα νέα κρατημέλη τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει στην έκθεση, όμως να φτιάξουμε και εδώ μια τροπολογία συμβαστική όσον αφορά τα θέματα της δυσκολίας των νέων κρατών μελών για να μπορέσουν να κάνουν την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων πλαισίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Άλφερ για τη βοήθειά του που είναι εμπειρογνώμος στο Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ επίσης και για τη βοήθεια από την γραμματεία, του συμβούλου, της ΙΤΡΕΒΕ. Ε, Περιμένω να ακούσω παρατηρήσεις και σχόλια από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Τώρα σας παρακαλέσω μισό μέχρι ένα λεπτό το πολύ ο καθένας. Κυρία Ριέρα Μαντού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα, σύντομα, για να υποστηρίξω και με την ομάδα μου τις περισσότερες από αυτές προτάσεις ε, της εισηγήτριας και για τις τροπολογίες των συναδέλφων σε σχέση με εκείνες επίσης της ομάδας μου και όπως εξήγησα προηγουμένως ε, γίνεται προσπάθεια να συμπληρωθούν όλα αυτά και να συμπληρωθεί ήδη η Πλήρη πρόταση τη κυρία Καρβάλια. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε για τι τροπολογίε ε, αυτέ. Ε, το έκανα σε προηγούμενη παρέμβασή μου για ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι κι αλλιώ οι συνάδελφοι που θα ε, παρέμβουν στη συνέχεια, το κάνουν επειδή εκείνοι τις έχουν συντάξει. Και για τις τροπολογίες από άλλες ομάδες, ε, συμφωνώ με την κυρία Καρβάλιο ότι είναι λίγες ε, αυτές οι τροπολογίες που θα έπρεπε να απομακρυνθούν, να απορριφθούν λίγες για θέματα που είναι εντελώς ξεχωριστά διαφορετικά από το θέμα αυτής της πρότασης. Είναι ε, θα πρέπει να δούμε ταυτόχρονα συμβιβαστικές προτάσεις ε, που θα πρέπει να είναι κάτι το περιληπτικό συνθετικό όλων αυτών. Είναι πολλά και σημαντικά που αναφέρονται εδώ. Και τελικό σχόλιο κύριε Πρόεδρε. Πεπισμένη είμαι ότι η επιτυχία, η ωφέλεια που θα βγει από αυτό ε, είναι επειδή στην Επιστημονική Επιτροπή αυτά που είπε έγιναν δεκτά και το RSE προωθήθηκε έτσι και γνωρίζουμε όλοι μας ε, ποια είναι αυτή η απάντηση για τον ακαδημαϊκό επιστημονικό κόσμο. Είναι εκείνοι άλλωστε που θα ωφεληθούν άμεσα από την εργασία μας. Ε, κυρία Καρβάλιο, να σας πω κάτι ειλικρινά, ότι το πετυχαίνουμε. Είναι η δική μου η άποψη που συμφωνεί με την άποψη επιστημόνων που συμφωνούν επίσης. Είναι συντονισμένη εργασία, καλή συνδυασμένη ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο οργανώσαμε ακροάσεις, επίσης διάφορες ε, συζητήσεις ε, με λεπτομέρειες συμμετείχαν και οι υπόλοιποι και επίσης αυτό το θέμα έχει σημασία μέσω σεμιναρίων και με την Ισπανική Προεδρία και τώρα τελευταία επίσης κατά τη διάρκεια της Βελγικής ε, Προεδρίας στο ξεκίνημα της η κυρία Καρβαλιό μπόρεσε να τα συλλέξει όλα αυτά, να τα συνδυάσει αυτές τις απαιτήσει, αυτές τις ιδέες, αυτές τις απόψεις στην εκθεσή της με ρεαλιστικό έξυπνο τρόπο και θα ήθελα και πάλι να τη συγχαρώ για αυτό που έκανε. Τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αγαπητοί συναδελφοί, υπενθυμίζω, εάν συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά θα συνεχιστεί η συνεδρίαση και το απόγευμα. Α, αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, κυρία Φόρτ. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια και για την προσέγγιση της και για την ακρόαση και για το ότι μας συμπεριέλαβε. Νομίζω πως οι λέξεις του εκπροσώπου της ΣΕΤΟ ήταν πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος απλοποίησης είναι να είμαστε σαφείς στο τι εννοούμε εξ αρχής και βέβαια ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους για να είναι οι συμβαστικές τροπολογίες σαφείς. Όταν μιλάμε τώρα για πρόθεση της αριστείας στην έρευνα που ακούστηκε τόσες φορές χτες και είναι το όραμα που χρειαζόμαστε. Όσον αφορά την ελαστικότητα και τη διατήρηση ελαστικότητας, μου άρεσαν τα σχόλια του Σουηδικού Πανεπιστημίου που μίλησε για την μέθοδο του πλήρους κόστους που τους βοηθάει και δεν θέλω να την χάσουν. Δεν άκουσα κανέναν ειδικό να ζητάει αύξηση του ανεκτού ποσοστού λάθους και αυτό είναι πολύ ευαίσθητο γιατί αυτό επιτρέπει ε, κάποια πράγματα. Δεν το ζήτησε αυτό, ζήτησαν απλοποίηση και να χρησιμοποιούν τις εθνικές λογιστικέ διαδικασίες. Και μήπω με την απλοποίηση αυτή μπορούμε να μειώσουμε τα σφάλματα και αυτό βεβαίως θα μας βοηθήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, για την εμπιστοσύνη. Αυτό, εντάξει, ισχύει για ορισμένους οργανισμούς, δηλαδή να δείξουμε εμπιστοσύνη και μιλάμε για λιγότερη διαχείριση, όταν μιλάμε όμως σε, για ιδιωτικό τομέα που με σκοπό το κέρδος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό μαζί με τον κύριο Κάρας εμείς είπαμε να δούμε πράγματα όπως ε, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή δάνεια και όχι επιχορηγήσεις. Οπότε να μην υπάρχει τόσο αυστηρή διαχείριση αλλά να υπάρχει ένας τρόπος διαχείρισης του ε, συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια παρένθεση. Ε, στην πρώτη μας αυτή συνεδρίαση εκπέμπεται μια πολύ ωραία εικόνα με τα μανίκια ανεβασμένα που σημαίνει ότι ξεκινάμε πολλή δουλειά αυτό το χρόνο. Για σας προσωπικά κύριε Πρόεδρε και μας δίνετε δύναμη ότι θα δουλέψουμε γερά. Ε, Ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια, ε, το κόμμα μας και μιλάω ως ε, το Ραπορτέρ εδώ. Ε, συμφωνεί με τις, τα σημεία της αναφοράς της κυρίας Καρβάλιο. Τρεις επισημάνσεις κύριε Πρόεδρε. Έχουμε κάνει μία πρόταση με τον κύριο Πουτικόφερ ως amendment για την διεθνοποίηση της συνεργασίας της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και ε, τεχνολογίας. Η δεύτερη, το δεύτερο amendment το οποίο έχω καταθέσει αναφέρεται στο Innovation Subgroup το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου στην ε, στο ραπόρτο της κυρίας Καρβάλιο και ήθελα να το τοποθετήσουμε εδώ υπενθυμίζοντας τις σοβαρές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως υποομάδα το Innovation Subgroup και η τρίτη δίνει έμφαση, η τροπολογία που έχω καταθέσει δίνει έμφαση στην ευρωπαϊκή ε, ε, περιοχή έρευνας. Αυτές είναι οι τρεις τροπολογίες οι οποίες από μας ε, υποβάλλονται για κάποια βελτίωση στο πολύ καλό κείμενο της κυρίας Καρβάλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ματίας, τον λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα προσπαθώ να να αποκριθώ στην εκκλησία σας να είμαστε σύντομοι. Ήδη αρκετές φορές είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και εδώ στην Επιτροπή αλλά και σε διάφορες ε, συναντήσεις που η συγγήτρια οργάνωσε. Σε δύο σχόλια θα ήθελα να προβώ. Καταρχήν ε, να προτείνω, να τονίσω τη σημασία αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας. Άλλωστε αυτό φάνηκε καθαρά και στις διάφορες συναντήσεις, αλλά και μέσω όσων και στο παρελθόν ασχολήθηκαν με την επιστημονική έρευνα. Εκτιμούν ακριβώς την αξία των προτάσεων ε, της εισηγήτριάς μας σίγουρα βελτιώνουν τα πράγματα και όσον αφορά την επιστημονική ας παραγωγή αλλά και την ποιότητα ζωής ε, όσων διεξάγουν αυτή την έρευνα και σχετικά με τις συμβαστικές προτάσεις ε, τροπολογίες της εισηγήτριας συμφωνώ με τις περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η σχετική διαδικασία προωθήθηκε παραδειγματικά γιατί κάλυψε πολλά και διάφορα και με τη βοήθεια όλων των ομάδων ε, δείξαμε ικανότητες σύγκλησης ε, να ακούσουμε ο ένας τις απόψεις του άλλου και να καταλήξουμε σε μία κοινή θέση, κάτι που νομίζω ότι πετύχαμε αν λάβουμε υπόψη μας τουλάχιστον όλα αυτά τα πράγματα και όσα υποστηρίζει ο καθένας. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά την εισηγήτρια για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο επετέλεσε την εργασία της. Νομίζω ότι έτσι εκφράζω και τις απόψεις των συναδέλφων που παρακολούσαν την διαδικασία. Ευχόμαστε να επανελειφθεί κάτι τέτοιο και στο μέλλον. Θα ήταν κάτι το πολύ καλό σαν σημείο σύγκλησης ανάμεσα σε αντιφατικές απόψεις. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους συναδελφούς τους Πένους. Ευχαριστώ την κυρία Καρβάγιο να αναφέρω έτσι επιγραμματικά τα σημαντικά για εμάς σημεία. Ο ενιαίος έλεγχος των βιβλίων που δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν θα πρέπει να υπάρχουν αλλαγές με αναδρομική ισχύ. Αν κάτι έχει πληρωθεί με ένα καθεστώς, δεν μπορεί μετά αναδρομικά η Κομισιόν να το αλλάζει. Δεν είναι πολύ άσχημο αυτό για τους ερευνητέ. Μετά θα πρέπει να δούμε τα καταποκοπήν ποσά και το τι γίνεται εκεί πέρα, να το συζητήσουμε και το αποφασιστικό βεβαίω είναι ο χρόνος μέχρι την εκταμίευση πρέπει να είναι συντομότερος. Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές που δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Νομίζω πως ε, παραμένει ανοιχτό το θέμα του ποια θα είναι μια καλή λύση για το ανεκτό ποσοστό σφάλματος όπου είναι βεβαίως διαφορετικά τα πράγματα στην έρευνα από ό,τι στα αγροτικά γιατί ε, εκεί πέρα πρέπει να είναι βεβαίως μικρότερο το ποσοστό ανεκτού λάθος γιατί είναι λιγότερο ποσοτικοποιήσιμα τα πράγματα στην ε, έρευνα αλλά βεβαίως είδαμε επίσης διότι γίνεται θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα ακόμα, τους φάρους, αν θέλετε. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ε, να υπάρξουν κάποια ορόσημα της ευρωπαϊκής έρευνας όπως το ΙΤΕΡ, παραδείγματος χάρη το οποίο αντί για ένα θετικό φάρος, ένα ορόσημο γίνεται τι να σου πω, ένα αρνητικό ορόσημο. Το Γαλιλαίο, παραδείγματο χάρη, θα ήταν κάτι στο, για το οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε υπερήφανοι. Είναι κάτι καλό, το υποστηρίζουμε όλοι, μέχρι και ο κύριο Τούρμα, το Γαλιλαίο τουλάχιστον. Και σε αυτά νομίζω πρέπει να εργαστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση και την ακρόαση χτες. Ε, αυτό το οποίο είδαμε είναι πως δεν μπορεί να υπάρχει μία μέθοδος και μία δικασία για όλους τους ε, τομείς. Ε, είναι αλλιώς ένα πανεπιστήμιο, ένα ερευνητικό ίδρυμα, μια, ένας μεγάλος όμιλος ή μια μικρή εταιρεία. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να έχουμε διαφορετικά σενάρια και βεβαίως το δεύτερο είναι ο ο χρόνος που πρέπει να γίνει μικρότερος όσον αφορά την εκταμείευση και παραδείγματο χάρη αν ε, μια επιχείρηση βιοτεχνολογίας ερευνά μια ασθένεια θα πρέπει να μπορεί να ε, εκταμιεύσει άμεσα τα λεφτά, αλλά δεν ξέρω βεβαίω. Είναι και οι κλίμακες χρονικές διαφορετικές. Ε, το ΙΤΡΕ αν έχει κρατήσει ή αν θα κρατήσει 50 χρόνια, αντιλαμβάνεστε πως είναι τελείως διαφορετικός ο χρόνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίστελ Ευχαριστώ και εγώ σύντομα, επειδή πιέζει ο χρόνος. Χτες στην ακρόαση είδαμε πως υπάρχει σοβαρή ανάγκη στην πράξη για να υπάρχει δυνατότητα επιλογής για εάν θα μιλήσουμε δηλαδή για καταποκοπή ποσά ή για το πώς θα καλυφθεί το κόστος. Και νομίζω σωστή ήταν η δήλωση της κυρίας Καρβάγιου στην αρχή πως ε, υπάρχουν και διαφορετικές ε, παραδόσεις και θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα και όχι τις ε, μεθόδους τις λογιστικές και βεβαίως δύο παρατηρήσεις ακόμα χτες προέκυψε πως χρειάζεται περισσότερη ευελιξία δυνατότητα προσαρμογής να λαμβάνουμε γρήγορα τις νέες πληροφορίες και βεβαίως όσον αφορά την αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού κανονισμού και την ψηφοφορία. Δεν πρέπει νομίζω να υποτιμάμε εδώ πέρα το τι θα γίνει με την Επιτροπή Ελέγχου. Εγώ είμαι, θα έλεγα πως θα πρέπει να αφιερώ, να, με συγχωρείτε, να βάσουμε το ανεκτό ποσοστό σφάλματος. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν ζήτησε σύντομα τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, σύντομη θα είμαστε. Και ευχαριστούμε την κυρία Καρβάλια και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας για το πόσο χρήσιμη και ενδιαφέρουσα είναι αυτή η έκθεση. Εκτός από τις ευχαριστίες θέλουμε να επαναλάβουμε την υπόσχεση του Γενικού Διευθυντή μας χθες στην ακρόαση που οργάνωσε η συγκεντρία ότι δηλαδή εμείς έχουμε δεσμευθεί. Θα λάβουμε διάφορα μέτρα για απλούστευση. Ορισμένα μέτρα θα είναι μακροπρόθεσμα, όμως ε, θέλουμε ακόμα και πριν την λήξη του νεστότος έτους κάτι να κάνουμε. Και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ κύριε Καρβαλιό. Θέλετε πάλι τον λόγο. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια. Σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που σχολίασαν και με βάση τα σχόλια που άκουσα σήμερα και τις διαβουλεύσεις και τις πολλές ακροάσεις και με τις δύο συνεδριάσεις που οργάνωσε η Βελγική και η Ισπανική Προεδρία θα είμαι σε καλή θέση να, προ... ευχάριστη θέση να προτείνω ε, κάποιες ε, συμβαστικές λύσεις και είτε αυτή την εβδομάδα και αύριο θα τα αποστείλω όλα αυτά και μετά θα έχουμε συνεδρίαση των ε, σκιωδών εισηγητών Στρασβούργο. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ απλά όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και τις προτάσεις τους. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Έχουμε τρία λεπτά για το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κυρία Τικάου, θα τα καταφέρουμε. Αλλιώ αναβάλλεται. Κύριε Τικάου. Ε, σε τρία λεπτά μπορούμε. Προσπαθήστε. Προσπαθήστε. Αλλιώς μια άλλη φορά. Γιατί ξέρω πως... Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το θέμα αυτό για τη Μαύρη Θάλασσα αξίζει μια συζήτηση για παραπάνω από τρία λεπτά. Ε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα και ελπίζω και οι συνάδελφοι να θελήσουν να συμμετάσχουν. Εδώ η στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα ξεκίνησε το 2007 και το 2008 δημοσιεύθηκε την Επιτροπή μια έκθεση. Εντάξει δεν μιλάμε για μια στρατηγική συγκεκριμένα, μια συνέργεια. Είναι η σύγκληση αρκετών πολιτικών κοινοτικών που εφαρμόζονται για τη Μαύρη Θάλασσα ενεργειακή πολιτική, παραδείγματο χάρη, πολιτική έρευνα επίση, ε, ε, γειτονίε, ε, εταιρική διεύρυνση μέσω τη Τουρκία και υπάρχουν διάφορε χώρε στην περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα με τι οποίε έχει εταιρική σχέση στρατηγική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ρωσία, όπως η Ουκρανία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τρεις τομείς την ενέργεια, την έρευνα και την βιομηχανική πολιτική. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι έχουμε Τρει εταιρικέ σχέσεις. Πρώτα απ' όλα ε, αυτή που ξεκίνησε το Μάρτιο φέτος για το ε, περιβάλλον, για την ενέργεια επίσης ε, και η Βουλγαρία είναι υπεύθυνη αρμόδια και μία ακόμα για τις μεταφορές με την Ελλάδα αρμόδια και υπεύθυνη. Σχετικά με τον ενεργειακό τομέα, θα πρέπει να πούμε ότι η περιοχή της ε, Μαύρης Θάλασσας έχει μία ξεχωριστή στρατηγική θέση επειδή είναι κοντά στην Κασπία. Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας παίζει σημαντικότατο ρόλο για την ενεργειακή ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την διαφεροποίηση όσον αφορά τις πηγές προμήθειας ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ακριβώς ε, αυτή την πτυχή όπως το σχέδιο Ναμπούκο που είναι πολύ σημαντικό ενεργειακά με δυνατότητα διαφοροποίησης των ε, πηγών προμήθειας ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μέσω και του κονδυλίων να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το σχέδιο. Ο διάδρομος ο Βόρειος είναι επίσης πολύ σημαντικός και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται να αναφερθώ και στο σχέδιο ΑΓΡΙ και στο σχέδιο ΠΕΟΠ e τα οποία θα μας επιτρέψουν ε, μια οργάνωση από ενεργικές πλευράς ώστε να ε, χρησιμοποιήσουμε τις πηγές εκεί ε, ενέργειας και να μεταφέρουμε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα να δούμε και την ε, έρευνα. Το 2009 αλλά και το 2011 θα έχουμε ένα σχέδιο για καλύτερη οργάνωση στην έρευνα για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας θα έχουμε 19 Ινστιτούτα ερευνητικά σε 6 χώρες που θα συμμετάσχουν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Να πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε μόλις ότι το δίκτυο Giant θα επεκταθεί και προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας οι χώρες αυτές θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην επιστημονική κοινότητα λοιπόν. Αυτά τα σχέδια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα έπρεπε κανονικά να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα αλλά μου δόθηκαν μόνο τρία λεπτά και δεν επαρκούν. Ίσως μετά από την ψηφοφορία οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να λάβουν το λόγο γιατί η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι τρομερά σημαντική για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντική γιατί έχει τομείς κλειδιά όπως μεταφορές, την ενέργεια, την έρευνα και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή αυτή. Να δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Οντί, ο οποίος ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ. Σύντομα, σύντομα να χαιρετήσω την εργασία του συναδέλφου και από το ξεκίνημα για το θέμα αυτό δεν είχε την πρέπουσα φιλοδοξία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2007 έχουμε αυτή την περιοχή μπροστά μας και με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία αυτή η συνέργεια έτσι σκέτη δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει να οθεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση για περισσότερη φιλοδοξία να επιδείξει για την περιοχή αυτή. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος δεν ζητάει τον λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν. Η έκθεση εξωτερικών θέλει να κάνει μια κρόαση και εμείς σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο για τον Σεπτέμβριο, οπότε έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση λοιπόν η οποία θα συνεχιστεί. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Α, η κυρία Τικάου πάλι. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σας είδα παρακαλώ. Ναι κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντι για όσα είπε. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή η περιοχή αυτή να, να γίνει αντικείμενο προσοχής και η ακρόαση με την Επιτροπή Ενέργειας το Σεπτέμβριο να δώσει κάτι το θετικό και περιμένω και τη συμμετοχή των συναδέλφων. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι μια περιοχή που νομίζω ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αλλά και την σταθερότητα στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στις ε, ψηφοφορίες. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση, ένα λεπτάκι. αν μπορώ να έχω λίγο την προσοχή σας. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω μια συνάδελφο η οποία έλειπε γιατί ήταν άρρωστη και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η κυρία Σισιλίκ επανήλθε και είναι ξανά μαζί μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Πιστέψτε με, ε, μας λείψατε σε πάρα πολλά ζητήματα και χαιρόμαστε που είστε ξανά μαζί μας. Όχι, ναι, πρέπει να το πω. Λοιπόν, περνάμε τώρα στις ε, τα σημαντικότερα τα είπαμε. Πρώτα απ' όλα, ψηφοφορία για τον προπολογισμό της κυρίας Χέρτσογκ είναι πολύπλοκη ε, υπόθεση. Ελπίζω να τα καταφέρουμε πρώτα απ' όλα όλες τις κάρτες. έχετε τις κάρτες της ε, ψηφοφορίας να τις δοκιμάσουμε λίγο Λοιπόν, ας ψηφίσουμε εάν ε, είστε ικανοποιημένοι που ξεκίνησε πάλι η δουλειά ή θα προτιμούσατε να είστε σε διακοπές. Άρχεται η θα προτιμουσετε να ειστε σε Πέρας. Ε, κάποιοι παραπάνω είναι εδώ μέσα. Ε, κάποιοι παραπάνω από το ΕΛΚ ψήφισαν υπέρ των διακοπών. Ναι, ναι. Τέσσερις παραπάνω από το ΕΛΚΑ, ένας πράσινος παραπάνω. Ε, Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας επίσης ένα παραπάνω. Οπότε, ξεκινάμε. Πρώτη ψηφοφορία. Να αναφέρω τα νούμερα, εάν μου επιτρέπετε, με τα δύο μόνο τελευταία ψηφία. 61-00 ε, κτλ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το 00 με προφορική τροπολογία Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 01 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 02 υπέρ. Κατά. Αποχές. 0,3 0-3 υπέρ. Κατά. Αποχές. 0,4 0-4 υπέρ. Κατά. Αποχές. 0,5 0-5 υπέρ. Κατά. Αποχές. 0,6 0-6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 07 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 08 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά έχουμε 68 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εποχές Εγκρίνεται. 61-72 ε, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Οπότε πάμε καταπίπτει. Πρέπει να ψηφίσουμε την 61-16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-20 και 68-15 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 21 και 68-16 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ταυτόσιμες πάλι 22 και 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 61-23 και 68-18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 61-81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 24 και 19 υπέρ κατά αποχές και αυτές εγκρίνονται ταυτόσιμες πάλι 26 και 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 61, 27 και 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 28 και 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Περνάμε τώρα στην 29 και στην 23 ταυτοσιμη υπέρ. Κατά Κατά εγκρίνονται. συγκρίνονται. ξανά 61, 30 και 68, 24 υπέρ. Κατά εποχε εγκρίνονται. 61, 31 και 68, 25 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνονται εγκρίνονται 61, 32 και 68, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 61, 33 και 68, 27 υπέρ κατά αποχές <coughs> εγκρίνονται 61, 34, 68, 28 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ναι να ψηφίσουμε μπλοκ. Όλη τη σελίδα αυτή. Καμία αντίρρηση να ψηφιστεί όλη αυτή η σελίδα μαζί από την 61-35 μέχρι 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και στην επόμενη σελίδα. 61-40 μέχρι την 37. Συμφωνείτε. Ψήφισμα αυτό το μπλοκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνεται. 68-31-1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 68-13 νούμερο 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Ερώτημα, να ξαναψήσουμε μπλοκ, όχι. Ε, 61-44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τις επόμενες μέχρι το τέλος της σελίδας μπορούμε να τις κάνουμε μπλοκ 47 δηλαδή μέχρι και 41 Μέχρι το 43, ωραία. Ε, ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνονται. Ήταν ταυτόσιμες. Περνάμε στην 61-53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να συνοψίσω πάλι κάποιες 56 μέχρι 59. Γίνεται. Αν μπλοκ. Ποιος είναι υπέρ αυτών των τεσσάρων. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 61-61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68-11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ με προφορική τροπολογία παρακαλώ Μπουτικόφερ κύριε πρόεδρε Θέλω να διαφωνήσω με την προφορική τροπολογία. Αυτό το οποίο προτείνεται εδώ πέρα έχει καλυφθεί ήδη από το ψήφισμα που έχουμε υιοθετήσει στο 08-05-01 στο 25 της κυρίας Χέρτσοκ νομίζω η ουσία καλύπτεται ήδη εκεί πέρα, γι' αυτό είμαι κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Ωραία, το λαμβάνουμε υπόψη, είναι κατά ο κύριος Μπιουτικόφερ, οπότε ψηφίζεται. Συμφωνούμε, καμία αντίρρηση. Ωραία, ψηφίζουμε την αρχική λοιπόν τροπολογία. Την 6182 χωρίς προφορική τροπολογία, ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ταυτόσημη. 76-77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 68 υπέρ. Κατά. Οπότε εγκρίνεται. Δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία περνάμε στην επόμενη. Συγχαρητήρια κυρία Χέρτσοκ, η οποία λείπει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν. Είναι δύσκολη αυτή η δουλειά. Περνάμε στην έκθεση Φανμπρέν. Περνάμε στην ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα η 24 η τροπολογία με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Τι, λάθος. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, λάθος. Ξέχασα την 4. Πρώτα απ' όλα η παρθμόν 4 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Όχι, 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Α, συγγνώμη, καταπίπτει, καταπίπτει, ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην 24 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 χωριστό τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική λύση 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπαριθμόν 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά να ξαναρωτήσω 43 υπέρ κατά ε, πρέπει να το ελέγξουμε, συγγνώμη. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι τρεις παραπάνω στο ΕΛΚ. Ένας πράσινος, δύο ΕΛΚ. Ε, το μηχάνημα το λέει. Τώρα τι να σου πω, λέει ψέματα. Είναι δυνατόν. Ε, κάποιοι άλλοι ψηφίζουν στους πράσινους τώρα εξακολουθεί να είναι ένας πράσινος. Ε, ευχαριστώ, αλλά... Ε, όχι, όχι κύριε Λάγκεν, όχι. Παρακαλώ αποσύρετε την, ε, την παρατήρησή σας, λέει η κύριε Λάγκεν, η οποία ήταν εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, εξακολουθούν να υπάρχουν παραπάνω βουλευτές. Μέχρι και ένας μείνει και όχι, ούτε τώρα. Ένα πράσινο παραπάνω, δύο η ευθύ ένας μη εγγεγραμμένο. Χαίρομαι που έρχονται εδώ πέρα οι συνάδελφοι στην ψηφοφορία. Μακάρι να συνεχιστεί και πέρα από αυτή την ψηφοφορία. Τρεις είμαστε. Ξέρω βεβαίως πως πολύ, ε, πολύ περισσότεροι να είμαστε εμπνεύματοι. Ε, ίσως η μηχανή να θεωρεί ότι είστε παραπάνω από όσοι πρέπει. Τι να πω, δεν, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έτσι, λέει ο πρόεδρος, λυπούμε. Μα δεν, δεν μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Τι θα κάνουμε. Έχω εδώ πέρα ένα κομπιούτερ μπροστά μου που μπορεί να κάνει και λάθος, αλλά μου λέει ένας πράσινος παραπάνω, δύο από την ε, Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας και ένα μη εγγεγραμμένο. Ή θα το λύσουμε τώρα ή θα κάτσουμε εδώ μέχρι αύριο. Λοιπόν, ξαναψηφίσουμε. Δεν ξέρω, εντάξει, ναι, μπορεί να έχει λάθος η μηχανή. Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, μηδενίστε το. Αρχίζει ξανά. Άρχισε η ψηφοφορία. Ναι, ναι, λύθηκε το πρόβλημα. Όχι, το ίδιο πρόβλημα. Ε, δεν, δεν μπορώ να αποφασίσω. Τι να σας πω. Είναι 54 έναντι 53. Λοιπόν, ο χειρός. Θα μετρήσει η γραμματεία. Σβήνουν όλα τα μηχανήματα. Παρακαλώ ποιο είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας. Υπέρ πρώτα. Ευχαριστώ κατά. Ε, αποχές. Κανείς, ωραία. 22 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται. Ελπίζω ε, να είναι σωστά η καταμέτρηση. Σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν συμβαστική παρισμών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ 45 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 53. Νέα προφορική τροπολογία ΕΚ. Ποιος θα την, θα την ε, διαβάσει. Είναι γραπτή η κυρία Φαν Θα τη διαβάσω. Νομίζω πως όλοι οι σκιώδεις τη γνωρίζουν. Είναι διαφορετική από αυτήν την οποία έχετε στον κατάλογο της ε, ψηφοφορίας και λέει όταν ψηθεί το σύστημα η... η ημερομηνία μεταξύ της αίτησης και της τελικής απόφασης δεν θα ξεπεράσει 4 με 6 μήνες ανάλογα με το τι έχει δώσει ο τελικός δικαιούχος. Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, οπότε ψηφίζουμε την 53 προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 54 υπέρ. Προφορική τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 καταπίπτει. 8 ε, του προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στα εκτιμώντας το υπαριθμό 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και συμβαστική 1 υπέρ όχι συγγνώμη 1 ε, του προπολογισμού πρώτα απ' όλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 του προπολογισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 και 18 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν πέρας 49 υπέρ 4 αποχές ένας δεν έχει κάρτα Οπότε νομίζω πέρασε. Ξεκάθαρα ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, την κυρία Φανμπρέντ. Οπότε τελείωσε αυτό το σημείο σχέση διάταξη. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 9, ενεργειακή στρατη... βιομηχανική πολιτική, με συγχωρείτε. Ο κύριος Λάγκε έχει το λόγο και μάλιστα μόνος του. Σας παρακαλώ να βγείτε ήσυχα από την αίθουσα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Kolleginnen, Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε μια νέα φρέσκια υφόρο βιομηχανική πολιτική και δύο πράγματα εδώ πέρα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο. Αφενός είναι σημαντικό να δούμε τη σημασία της βιομηχανίας για τη δημιουργία πλούτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την εξής κατάσταση. Τρία, τρία τέταρτα των εξαγώνων βιομηχανικά προϊόντα. 25% του ΑΕΠ παράγεται από τη βιομηχανία. Παρόλα αυτά, συχνά υπάρχουν απόψεις πως είναι κάτι το παλιό και βρώμικο η βιομηχανία. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε νέα, μια νέα φρέσκια βιομηχανική πολιτική. Ακριβώς ειδικά όταν μιλάμε για την διαδικασία ανανέωσης που περνάει η βιομηχανία. Και βεβαίως το η δεύτερη εποδός την οποία πρέπει να λαμβάνουμε είναι πως η βιομηχανική βάση πρέπει να διατηρηθεί στην Ένωση και αυτό σημαίνει βεβαίως και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας που μιλάμε για πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία οπότε νομίζω σωστό είναι τώρα να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και να έχουμε μια νέα φρέσκια βιομηχανική πολιτική γιατί βεβαίως έχουμε και νέες προκλήσεις ε, που προδιαγράφονται τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως έχουμε την πίεση της παγκοσμιοποίησης, ενώ σε άλλες χώρες έχουμε νέες αγορές και γίνονται και νέες επενδύσεις. Οπότε νομίζω η δυνατότητα της καινοτομίας θα ενισχυθεί για να υπάρξει κάποιος ανταγωνισμός και νομίζω για τη στρατηγική του κόστους δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό με τη μείωση κόστου. Πρέπει να είμαστε ηγέτε στην τεχνολογία για να μπορούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Βεβαίω, αντίθετο ζήτημα, πως έχουμε και οικολογικές ε, προκλήσεις. Εάν το πάρουμε στα σοβαρά να παραμείνουμε εντός των δύο βαθμών, τότε θα πρέπει η βιομηχανική βάση να ανανεωθεί, να χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους για να έχουμε λιγότερες εκπομπές. Και βεβαίως νέα επιχειρηματικά παιδεία ακριβώς για να παράγουμε σεβόμενοι το κλίμα. Και η τρίτη πρόκληση, το θέμα των δημογραφικών εξελίξεων που είναι ήδη πρόβλημα στην αγορά εργασίας για να βρεθούν ε, άτομα που θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα και αν γερνάμε και όλοι μαζί νομίζω θα ενταθεί το πρόβλημα αυτό αλλά θα έχουμε και διαφορετική κοινωνική δομή η οποία απαιτεί νέες διαδικασίες παραγωγής και νέα προϊόντα και αυτό είναι σοβαρή πρόκληση οπότε από την εποδό αυτή που ανέφερα και την πρόκληση που πρέπει να έχουμε κατά νου πρέπει να δούμε το νέο ορισμό της βιομηχανικής πολιτικής όπως γνωρίζετε η Κομισιόν έκανε κάποιες πρώτες σκέψεις στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 και ξεκίνησε κάποιες ε, πρωτοβουλίες ορόσημα και αναμένουμε στις 13 Οκτωβρίου τις προτάσεις της Κομισιόν για να προσπαθήσουμε από κοινού να τοποθετηθούμε. Νομίζω πως ο νέος ορισμός μηχανικής πολιτικής απαιτεί να φύγουμε από την άμεση πολιτική των παρεμβάσεων αλλά νομίζω πως πρέπει να φύγουμε και από την πολιτική που λέει μόνο εμείς δημιουργούμε το πλαίσιο και όλα τα άλλα τα κάνει η αγορά. Οπότε προσπάθησα στο έγγραφο αυτό εργασίας να σκιαγραφίσω μια πολιτική βιομηχανική που έχει ένα οριζόντιο επίπεδο που διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αλλά και μια τομεακή διάσταση για κάποιους κλάδους ε, της βιομηχανίας. Εάν δούμε λοιπόν το οριζόντιο επίπεδο, βεβαίως μιλάμε για μια αλυσίδα καινοτομίας που πρέπει να προωθηθεί για την απλοποίηση του προγράμματος πλαισίου πρέπει λοιπόν να έχουμε σε όλα αυτά τα κομμάτια της ε, αλυσίδας καινοτομία για την βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη μια καλύτερη οργάνωση. Δεύτερον, βεβαίως, το θέμα είναι η βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε το ότι η παραγωγικότητα της εργασίας έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά η, παραγωγική χρήση των πόρων δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ Γι' αυτό θεωρώ πως ειδικά εάν είναι να έχουμε τεχνολογική ηγεσία θα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό και πρέπει να έχουμε και βεβαίως κατάλληλους δίκτες και λογικούς δείκτες και θα πρέπει να μετρήσουν οι επιχειρήσεις την αποτελεσματική χρήση των πόρων και να τη βελτιώσουν. Επίσης, εδώ πέρα μιλάμε και για τις πρώτες ύλες, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες αυτό συζητιέται, το θέμα των εξ, της εξωτερικής προμήθειας πρώτων υλών. Έχουμε έντονους ανταγωνιστές. Και μιλάμε πια για μονοπόλιο στην αγορά πρώτων υλών ειδικά όσον αφορά κάποια μεταλλεύματα έχουμε τρεις εταιρείε που μονοπολούν 75% ε, της αγοράς οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για τους προμηθευτές των πρώτων υλών αλλά και να δούμε τι κάνουμε με τις πρώτες ύλες και πρέπει νομίζω να οδηγηθούμε σε έναν κύκλο ανακύκλωσης και βεβαίω οι πρωτοσύλλες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Να υπάρξει δηλαδή και μια γεωγραφική τράπεζα και γεωλογική τράπεζα δεδομένων για να ξέρουμε πού βρίσκεται τι. Το θέμα της ενέργειας. Η υποδιπλή έννοια είναι σημαντικό αφενός επαρκή ενέργεια χρειάζεται η βιομηχανία και βεβαίως από την άλλη να υπάρχει υπό μορφή ώστε να προστατεύει το κλίμα και να δημιουργήσει έτσι νέες θέσεις εργασίας. Και, και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και βεβαίως θα υπάρξει μια αναδιάρθρωση που θα πρέπει να την συνοδεύσουμε. Σαφέ, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε όλες τι βιομηχανικέ δομέ. Μια φορά έχουμε ε, την εξή κατάσταση κάνουμε τους πυροσβέστες όταν κάτι διαλύεται ε, ίσως να επεμβαίνουμε πάρα πολύ αργά στην εξέλιξη του άνθρακα και του χάλιβα αναπτύξαμε τέτοιες πολιτικές, ε, κοινωνικές πολιτικές και θα πρέπει να ε, τις ενισχύσουμε αυτές έτσι ώστε να μην ε, παρατηρούμε μόνο τη διαδικασία όταν έχει γίνει η ζημιά αλλά να προσπαθούμε να έχουμε αυτή τη μετάβαση από τις παλαιές στις νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό θα γίνει και με τα διαρθρωτικά ταμεία και με το Ταμείο της παγκοσμιοποίηση προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Για να δούμε και το θέμα των προσόντων που είναι πάρα πολύ κεντρικό σε όλα τα, τα επίπεδα. Ε, ειδικά όσον αφορά τα προσόντα υψηλού επίπεδου. Και εδώ πέρα υπάρχει την έννοια, η έννοια βεβαίως της παραδοσιακής εκπαίδευσης και της ε, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ε, και η διαδικασία Μπολόνια 2. Αυτές νομίζω είναι κάποιες πτυχές του οριζοντίου επίπεδου και επιπλέον ε, έχουμε και κάποιες προτάσεις για τις τομεακές δραστηριότητες που αναφέρονται στο έγγραφο εργασίας, ειδικά στους κλασικούς τομείς, ε, αυτοκίνητα, ναυπηγεία, χάλιβας, αλλά και τους νέους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη, ε, αιωλική ενέργεια και εκεί πέρα απαιτείται μια τομεακή αντιμετώπιση και όπως έχουν πάει τα πράγματα τώρα με το CARS 21 και την ομάδα δράσης υψηλού επίπεδου θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε πιο δεσμευτικούς στόχους και να δούμε τι θα γίνει και στην εφαρμογή. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε δει το έγγραφο εργασία με, με τις 15 προτάσεις μου και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Τέλος, μία πτυχή ακόμα. Πιστεύω πως η πολιτική θα είναι επιτυχής μόνο αν υπάρχει μια ενσωμάτωση, μια ολοκλήρωση. Εγώ έχω την αίσθηση πως αυτό δεν, τυχαίνει πάντα στην, ε, δεν πετυχαίνει πάντα στην Κομισιόν. Έχουμε δηλαδή μια ψηφιακή ευρωπαϊκή προοπτική, μετά μια περιβαλλοντική πτυχή, μια βιομηχανική πτυχή και στην Κομισιόν πρέπει να τα δουν όλα αυτά μαζί, αλλά και μεταξύ ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτικής των κρατών μελών πρέπει να υπάρξει συντονισμό. Το άρθρο 173 δηλαδή πρέπει να ενεργοποιηθεί, αλλιώ πλέον δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε. Αυτά και σα ευχαριστώ και αναμένω τα σχολεία σας. Ευχαριστώ αυτές συνάδελφε. Να υπενθυμίσω 11 και 30 θα έρθουν οι Βέλγοι Υπουργοί με δύο, πράγμα, δύο σημεία τη ημερήσια διάταξη πρέπει να έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, οπότε 11 η ώρα θα ασχοληθούμε με το επόμενο θέμα. Γι' αυτό το σημείο λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε ζητήσει 10 τον λόγο. Αυτό σημαίνει πω θα παρακαλέσω όλου του συναδέλφου να είναι σύντομοι. Πρώτα απ' όλα η κυρία Γκροστέτη της Κιώδης, συγγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Με προσοχή διάβασα το έγγραφο εργασία του εισηγητή μα και τι διαπίστωσα η νέα προσέγγιση για τη βιομηχανία στην Ευρώπη πηγαίνει βάσει 15 σημείων κλειδιών. Φοβάμαι κάπως ε, ότι έχουμε ένα κατάλογο ευχών, πόθων ε, και ότι θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Κρίμα θα ήταν πάντως ε, για μια τόσο σημαντική έκθεση θεμελιώδους σημασίας. Ε, θα πρέπει να προσφέρουμε απαντήσεις στην κρίση. Ε, σε τρεις άξονες να βασίσω την στάση μου. Πρώτα απ' όλα οι ευρωπαϊκές μηχανίες να αξιοποιηθούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει ποιε είναι οι προτεραιότητες, εκεί να εστιάσουμε με τα τεχνολογικά προγράμματα μακρόπνοα Υπάρχει βέβαια ανάγκη να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια να δούμε και τις κατευθύνες γραμμές σε ορισμένους άξονες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Μίλησε για αυτά ταχιστά ο εισηγητή. πρώτα απ' όλα για την προσέγγιση που θα πρέπει να έχουμε, τομεακή οριζόντια, είναι σημαντικά και τα δύο και διάφορα κοινά που θα επηρεάσουν ιδιαίτερα αρκετού τομεί οριζόντια προσέγγιση αυτή και επίσης ιδιαίτερα να προσέξουμε τα μεγάλα σχέδια, αυτή είναι η τομεακή προσέγγιση. Οι εταίροι μας αλλά και οι ανταγωνιστές μας σε παγκόσμιο επίπεδο το ίδιο κάνουν ε, και στα πλαίσια της Αμερικής στρατηγικής για την καινοτομία η στρατηγική αυτή που ακολουθήθηκε, υιοθετήθηκε τον Αύγουστο του 2009 από τον πρόεδρο Ομπάμα ε, καθορίστηκαν εκεί τομεακές προτεραιότητες ας πούμε για τα καθαρά αυτοκίνητα ή τα για την υγεία το ε, τομεακά. Χρειάζεται, απαιτείται μια χρηματοδότηση όπως τόνισε και ο εισήγητης ε, το PCRD. Εκεί θα πρέπει να το προσέξουμε, θα πρέπει να δούμε τα κονδύλια πώς δεν θα αυξηθούν, να δούμε ποιες ε, θα είναι προτεραιότητές μας, όπως θα τις καθαρίσουμε και χρησιμοποίηση των εργαλείων αυτών των οικονομικών. Να έχουμε πρόσβαση επίσης κεφάλαια κινδύνου, δεν θα πρέπει να το, να το φοβόμαστε αυτό. Επίσης διάφορα μεγάλα σχέδια και επίσης και να δούμε. Σημαντικό είναι από τη στιγμή που μιλάμε για καινοτομία. Χρειάζεται να προσέχουμε. Δεν θα πρέπει να προσέχουμε μόνο την καινοτομία. Η παραδοσιακή βιομηχανία με πάρα πολλές θέσεις εργασίας, το τόνισε ο εισηγητής, ε, θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η βιομηχανία, να προστατευθεί η καινοτομία να γίνει παραγωγή μόνο μέσω μιας παραδοσιακής ισχυρής βιομηχανίας που να είναι πάντα εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι συμπληρωματικά λοιπόν και τώρα η καινοτομία για την ε, ανταγωνιστικότητα των μηχανιών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει ελκυστική, να είναι ελκυστική, να αποφύγουμε επιβαρύνσεις και περιπλοκές εδώ μπερδέματα στην όλη οργάνωση, σε όλους αυτούς τους τομείς. Διαθέτουμε πολιτικές, μιλάμε για την ελάφρυση των διοικητικών ε, βαρών, αλλά δεν θα πρέπει μόνο να το συζητάμε, χρειάζεται να είμαστε και αποτελεσματικότεροι, πολύ πιο αποτελεσματικοί από ό,τι σήμερα. Να δούμε την καινοτομία που δεν είναι μόνο τεχνολογικής φύσεως, είναι δημιουργικότητα, είναι το marketing, είναι το design και σαν πάρα πολλούς τομείς που δεν είναι τεχνολογικοί μια υπενθύμηση. Χρειάζεται να επαγρυπνούμε, το τόνισε ο εισηγητής, να υπάρξει μια ψηλότατο επίπεδο κατάρτιση εκπαίδευση. Χρειάζεται να το στηρίξουμε αυτό, την εκπαίδευση αυτή. Τρίτο σημείο και ολοκληρώνω να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω μιας ευάθης στην εσωτερική αγορά και με μια εξωτερική πολιτική με ιδιαίτερο σθένος και με ένα καλό, σωστό ανταγωνισμό, όχι στρεβλωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην θίξουμε του υπάρχοντε ισχύοντε κανόνε, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι κάνουν σε διεθνέ επίπεδο οι ανταγωνιστέ μα. Να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε καλύτερα σε αυτό που κάνουν, να μην σκεφτόμαστε μόνο στα στενά πλαίσια των συνόρων μα. Δεν είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο η Ευρώπη που θα ελεγχόταν ε, τα κρατικά κονδύλια. Ε, θα μπορούσαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην μας φεύγουν οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις, να μην υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού, χρειάζεται να εξετάζουμε τι γίνεται και αλλού και γιατί όχι και εμείς τα ίδια να κάνουμε όπως και οι υπόλοιποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν πετύχει την άρση των εμποδίων σε, ε, ε, στις, και στις δημόσιες αγορές, θα πρέπει να δούμε τότε πώς θα υπάρξουν αμοιβαία μέτρα που θα ισχύσουν και για το περιβάλλον επίσης ε, χρειάζεται αυτό να το συλλογιστούμε. Είναι και γνώση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δικό μας θέμα εσωτερικό. Χρειάζεται αυτό να, το, να προχωρήσουμε σε εξαγωγές αυτής της γνώσης ποιοτικής παραγωγής, την ποιοτική μας παραγωγή ακριβώς. Ε, γιατί αν δεν μπορέσουμε, αν δεν ξέρουμε να πουλήσουμε αυτό που ξέρουμε, οι άλλοι δυστυχώς γνωρίζουν αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι άλλο. Στην πρόσβαση στις πρώτες είπε γι' αυτό ο εισηγητής, είναι σημαντικό και προσδιορίσε η Επιτροπή 14 πρώτες ε, που έχουν ιδιαίτερη σημασία και τα 20 επόμενα χρόνια θα τριπλασιαστεί η κατανάλωσή τους. Και με το ανάπτυξη της πράσινη τεχνολογίας σε λίγες χώρες υπάρχουν. Κίνα, Βραζιλία, στο Κονγκό που περιορίζουν όμως την, ε, το εμπόριό της αυτά και θα πρέπει να δούμε και στα πλαίσια του ΠΟΕ τι μπορεί να γίνει και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την πολιτική μας ε, για να χρησιμοποιούμε τα απορρίμματά μας μπορούμε έτσι να αντισταθμίσουμε και την έλλειψή μας σε παρόμοια υλικά. Ολοκληρώνω, τάχιστα κύριε Πρόεδρε, να μην ξεχνάμε και όσα μας απασχολούν για το περιβάλλον στα πλαίσια μιας πράσινης οικονομίας και να έτσι και όσα μας απασχολούν να τα εκφράζουμε μέσα των αποφάσεών μας, αλλά ταυτόχρονα αυτές να μπορούν τις αποφάσεις να τις αντέξουν και οι εταιρείε μας, οι βιομηχανίε μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, ευχαριστώ. Να πω πως η κυρία Γκροστέτ ε, νομίζω μπορεί να μιλήσει και καλύτερα από τον κύριο Λάγκε από την ε, τον κύριο Λάγκεν, γιατί στη Γαλλία έχουν εδώ και χρόνια βιομηχανική πολιτική, καλύτερη από ό,τι υπήρχε στη Βρετανία ή στη Γερμανία. Αλλά αυτές οι υποτιθέμενες βρώμικες επιχειρήσεις ε, δεν θα πρέπει να τις αποφεύγουμε. Πρέπει να πούμε πως ε, είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτές. Τώρα, ναι, χρειαζόμαστε αηφόρο εξέλιξη της ε, βιομηχανικής βάσης, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται βεβαίως και αλλαγή των χρηματαγορών και εδώ πέρα είναι το σημαντικό η καινοτομία. Επίση. τώρα εγώ το βλέπω κάπως πιο επικριτικά. Δεν θα πρέπει να είμαστε ρυθμιστικοί και προστατευτικοί. Εντάξει, μπορούμε να τα δούμε από την πλευρά του ανταγωνισμού. Έχουμε καλά προϊόντα, π.χ. στον τομέα των αυτοκινήτων, όπου σε κάποιου τομεί έχουμε πάνω από 80% της παγκόσμιας παραγωγή. Δεν χρειάζεται προστατευσμό, χρειάζονται μόνο καλά προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πως οι δυνάμει της αγοράς μας δείχνουν τον δρόμο προς την καλύτερη τεχνολογία. Γιατί τι βλέπουμε εδώ πέρα. Κάνουμε εμεί διατάξει που είναι πάρα πολύ λεπτομερεί ότι χρειαζόμαστε μέχρι το τότε, το 2015, 38,4 μείωση των εκπομπών. Ε, δεν ανάγκη τόση λεπτομέρεια, πρέπει να δούμε απλά οι καλύτερες τεχνολογίες να εφαρμόζονται και από τις δυνάμεις αγοράς. Η κυρία Γκροστέτ τώρα είπε πως ε, η πρόθεση της έρευνας είναι μεγάλο κομμάτι. Αυτό θα γίνει όμως εάν μπορούμε να προωθήσουμε και την καινοτομία για να μπορούμε να πουλήσουμε κάτι το οποίο θα είναι καινοτόμο οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε στο πλαίσιο του 7 πλαισίου έρευνας αηφορία κύριε Λάγκε συμφωνώ συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι ε, ένα από τα βασικά και ε, συνεχή της ε, βιομηχανικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας, ε, καλύτερη αποτελεσματικότητα. Οπότε η βιομηχανική ε, προσέγγιση εδώ πέρα είναι αυτή η οποία χρειάζεται. Επίσης, λέτε πως δεν θα πρέπει να κάνουμε λιγότερους κανόνες και ίσως περισσότερες καμπάνιες Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε ίσω καμπάνιε και λιγότερου κανόνε κάποιε κάποιες για να βελτιώσουμε νομίζω και να επηρεάσουμε καλύτερα τι αγορέ. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω πρέπει να αφήσουμε εκτό τη μικρή βιομηχανία, ειδικά να μην του επιβαρύνουμε με αυτέ τι υποχρεώσει εκθέσεων και γραφειοκρατία και να αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πέσουν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια. Συμφωνώ πλήρω με την κυρία Γκροστέτ όταν μιλάει για το Made in πρέπει να επιμείνουμε στα προϊόντα μας. Είμαστε ένας από τους λίγους παγκόσμιους χώρους που δεν έχουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Οι Αμερικανοί έχουν απέτηση να λένε από πού προέρχεται το προϊόν. Οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, εμείς, το ίδιο, εμείς δεν έχουμε. Λάθος. Γι' αυτό είμαι υπέρ του Made in. Τελευταίο, πρέπει να είμαστε υπέρ των προϊόντων ε, σημεών, εάν θέλετε, για να μπορεί να πείσει και η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Παραδείγματο χάρη Airbus. Με το Airbus τα καταφέραμε στη, να θέσουμε τους κανόνες στην παγκόσμια αγορά και να περάσουμε και πρώτοι. Τέλος. πρέπει να τα πούμε αυτά και στους πολίτες μας α, ως πολιτικοί. Να έρθουμε σε ένα διάλογο με τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα πως το έγγραφο αυτό του κυρίου Λάγκεν είναι μια καλή βάση συζήτησης, ε, αναφέρει πάρα πολλές πτυχές και αυτό είναι αναγκαίο και σωστό. Πράγματι η βιομηχανική πολιτική, εάν την παίρνουμε τόσο σοβαρά όσο μας ο κύριος Λάγκε, δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν είμαστε πολύ στενά στοχευμένοι, γιατί υπάρχουν κάποιες κοινωνικές συνθήκες για το εάν πραγματικά λειτουργεί η βιομηχανική πολιτική και έτσι αντιλαμβάνομαι ε, την προσέγγισή σας ότι θέλετε να τα δείτε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να ε, φτάσει η συζήτηση να καταλήξει σε ένα υπόδειγμα, σε ένα όραμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θεωρώ επίσης πως αυτό δεν είναι κάτι το περιττό γιατί θα συνεισφέρει στο να γίνει μια συνολική προσπάθεια από όλη την κοινωνία για να εφαρμοστεί δεν είμαι σίγουρος, ε, κύριε Κωστέτο, ότι σας άκουσα καλά, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να θεωρήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική ως μίμηση άλλων και ότι αν κάποιοι κάνουν κάτι άλλο εμείς θα τους ακολουθήσουμε. Όχι, εγώ θα ήμουν υπερήφανος ε, να έχουμε μόνο ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, να μην ακολουθούμε τους άλλους εμείς οι ίδιοι να ανοίγουμε νέους δρόμους. Δύο, ε, σε δύο πράγματα δεν είμαι σίγουρος ε, κύριε Λάγκε ε, ότι τα βλέπουμε τα πράγματα ακριβώς ίδια. Το πρώτον, η σχέση της βιομηχανικής πολιτικής με την παγκόσμια τοποθέτηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ήδη είναι παγκόσμια. Η μεγαλύτερη επένδυση της BASF, παραδείγματος χάρη, είναι στην Κίνα. Και αυτή η επιχείρηση βεβαίως θεωρεί αυτόν ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια. Οπότε, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει παγκόσμια θέση των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να ε, ορίσουμε και το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το δεύτερο σε σχέση με μια συνεκτική και σαφή βιομηχανική πολιτική αναφέρθηκε από τον κύριο Χατζημαρκάκη πως υπάρχουν διαφορετικές εθνικές παραδόσεις και δεν είμαι σίγουρος πως ε, με ένα μεγάλο άλμα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Γι' αυτό εγώ λέω να επικεντρωθούμε σε κάποια κεντρικά ζητήματα Οπότε το να λέμε πως οι δυνάμεις ε, της αγοράς θα εφαρμόσει την καλύτερη τεχνολογία μου φαίνεται λίγο αισιόδοξη. Άλλοι την, ε, θεωρούν την ε, πυρηνική ενέργεια την καλύτερη. Ε, ναι, αλλά χωρίς επιδοτήσεις δεν θα πήγαινε πουθενά. Οπότε μη λέμε μόνο ότι είμαστε κατά τους, ε, του κράτους και παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα στο θέμα της καινοτομίας. Το υποστηρίζω, όπως και η κυρία Γκροστέτ, αυτή την ευρύτατη προσέγγιση και καλό είναι να μιλήσουμε για ανθρωποκεντρική καινοτομία και να δούμε το ζήτημα της αξιολόγησης της τεχνολογίας. Σημαντικό επίσης είναι η έμφαση στην αποτελεσματικότητα των πόρων, την οποία εγώ θα ήθελα να μετρήσω στα προϊόντα και όχι στο επίπεδο της εταιρεία. δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα, αλλά να περάσω στο θέμα των πρώτων υλών. Κατά την απόψή μου πρέπει να υπάρχει και μια διαφάνεια των αγορών. Η Γαλλία ήδη έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, π.χ. το σιδηρομετάλλευμα συσσωρεύεται για να γίνει μετά κερδοσκοπία. Είναι βασικό κομμάτι λοιπόν της ευρωπαϊκής πολιτικής αυτό. Και πρέπει να δούμε βέβαια την σχέση της εμπορικής πολιτικής με τη βιομηχανική πολιτική. Στο παρελθόν κάναμε βιομηχανική πολιτική μέσω της εμπορικής ε, πολιτικής. Αυτό είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Και τέλος, στο σημείο 13 που το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό με τους όρους αυτούς πράγματι πρέπει να μιλήσουμε για την κατάσταση των νέων γιατί είναι πάρα πολύ υψηλή ανεργία να δούμε το θέμα των γυρεωτέρων και τρίτον την κατάσταση όσον αφορά τους μηχανικούς στο Ροστόκ ε, πρόσφατα ξεκίνησε ένα, νέα, ένα νέο εργοστάσιο της εταιρείας Σούσλον, μιας Ινδικής εταιρείας που φτιάχνει ανεμογεννήτριας. Ο δε διευθυντής είπε πως ε, πάμε στη Γερμανία γιατί εκτιμούμε τους Γερμανούς μηχανικούς. Αλλά εάν ε, εμείς εισάγουμε Ινδούς μηχανικούς ε, την πατήσαμε. Οπότε πρέπει να δούμε και το ζήτημα της εκπαίδευσης των μηχανικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση για να ασχοληθούμε και με τα άλλα θέματα, αλλά έχουμε ακόμα 10 άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, τι να κάνω τώρα. Σας ρωτάω εσάς. Ε, σας παρακαλώ, ε, δεν ξέρω αν κάποιος δεν θα ήθελε να μιλήσει και κάποιος άλλος να μιλήσει μόνο μισό λεπτάκι. Ε, εντάξει, ε, να δώσω άλλα έξι λεπτά. Αλλά, εντάξει, πρέπει να ε, συζητήσουμε και την άλλη έκθεση και 11.30 ώρα λυπούμε, ε, έρχονται οι υπουργοί. Άντε να περιμένουν πέντε λεπτά, όχι μισή ώρα. Ή μπορούμε να συνεχίσουμε και ό,τι γίνει. Και ο καθένας να μιλήσει όσο θέλει και ξαναρχόμαστε το απόγευμα. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να είστε λίγο πειθαρχημένοι. Ε, επί της διαδικασίας, αν θέλετε, μόνο μία σύντομη πρόταση. Να μιλήσουν οι σκιώδεις. Ναι, ναι, οι σκιώδεις θα μιλήσουν. Νομίζω μίλησαν όλοι οι σκιώδεις, λέει ο πρόεδρος. Όχι, τη Γκουε δεν μίλησε, λέει ο κύριος Τούρμες. Όλοι, όλοι οι σκιώδεις μου είπαν. Λοιπόν, ωραία, οι σκιώδεις, σωστό. Κύριε Πρόεδρε, θα στείλω γραπτό στην παρέμβασή μου και επίση με ηλεκτρονική διαδρομή σε όλου του βουλευτέ, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Υπάρχουν ορισμένοι που μιλάνε για 10 λεπτά και άλλοι δεν μπορούν να βγάλουν κουβέντα. Τι γίνεται. Θα πρέπει να το οργανώσουμε, ώστε όλε οι ομάδε να παρεμβαίνουν τρίτη φορά που εμείς οι νοτικές τώρα δεν μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να οργανωθούμε ε, τι θα κάνουμε ακριβώς. Εντάξει, δεν θα μιλήσω, θα σας τη στείλω γραπτός. Όχι, όχι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, όχι, τώρα θα μιλήσει η κάθε ομάδα, η κάθε ομάδα, αυτό είναι το σημαντικό, αυτό θα κάνουμε και μετά βλέπουμε. Συμφωνώ. Λοιπόν, ε, βοηθήστε με και εσείς λίγο. Λοιπόν, οι ομάδες μίλησαν, μίλησαν. Λοιπόν, Ντεχέν λοιπόν. Γιατί δεν μίλησε ακόμα η ομάδα σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γρήγορα αλλά θα είναι δύσκολο. Εδώ η απασχόληση, η βιομηχανία, όλα αυτά μετά από την τελευταία κρίση. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Ίσως να ντύσουμε το χάπι το πικρό με σοκολάτα για να γλυκάνει. Υπάρχουν πράγματα που δεν εξετάζονται σημαντικά, αλλά εξετάζονται βιομηχανία που θα σέβεται περισσότερο το περιβάλλον. Αυτό σοβαρά αντιμετωπίζεται. Τίποτα μας για την κοινωνική πτυχή. Έτσι, αυτό το καρκίνο που διαβρώνει τη βιομηχανία και για τη πίεση της Ευρώπης αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται από από μια αιστεία που αφορά μόνο την ωφελημότητα και ε, μόνο και μόνο οι μέτοχοι για να έχουν μερίσματα υψηλότερα αυτούς, αυτοί ικανοποιούνται. Εδώ και επίσης οι αναδυόμενες οικονομίες εποφελούνται. Εδώ κοντά στο σπίτι το δικό μου υπάρχει μια ειδικευμένη βιομηχανία με φίλτρα για την βιομηχανία την πυρηνική έκλεισε γιατί οι Αμερικανοί την αγόρασαν την εταιρεία και πήραν ε, τις άδειες εκμετάλλευσης και έφυγαν την έκλεισαν. Εντάξει, υπάρχει αυτή η διάφραση από αυτό το ντρομερό καρκίνο της μόνιμης αναζήτησης κέρδους. Θα πρέπει να έχουμε την πολιτική, τη βιομηχανική του θάρρους ε, για να σπάσουμε αυτήν την αλυσίδα για μια βιομηχανία που θα βασίζεται στην ανάγκη να ανταποκριθεί κανείς στις ανάγκες του πληθυσμού μας. Ε, ναι, για να πούμε ναι, ναι σε μια βιομηχανική κοινή πολιτική πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού μας, ναι σε κοινή βιομηχανική πολιτική που θα σέβεται το περιβάλλον με λιγότερη ενέργεια που θα απαιτείται και λιγότερες ύλε, ναι σε μια βιομηχανική κοινή πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη της την απαραίτητη ανάπτυξη όλου του χώρου. Ναι, όταν σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων και ένα καθεστώς κοινωνικό που θα είναι άξιο του όνοματός του και ναι, όλα αυτά που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν οικονομικά όλες οι χώρες, όλη η Ευρώπη. Βέβαια όλα αυτά είναι κατά το συμφέρον της αγοράς και κυρίως κατά του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Ας δειχτούμε τρελή, ας τροποποιήσουμε τον καταστατικό της Ευρώπης. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω πως η Επιτροπή μας πρέπει να συζητήσει περισσότερο το τι θα κάνουμε και να στηρίξουμε στρατηγικά τη βιομηχανική πολιτική στο μέλλον. Και η κρίση έδειξε πως η αξιοπιστία και η φερεγγιότητα και η ρευστότητα των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική και τώρα με την εξυγίανση των χρηματοοικονομικών βεβαίως πάλι το βασικό βάρος θα το σηκώσει η βιομηχανική πολιτική και η μείωση βλέπετε η πίεση των μισθών. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα τον κύριο Λάγκε γιατί ανέφερε την ίση μεταχείριση στη φορολογία και νομίζω στο παγκόσμιο πλαίσιο εάν δείτε το τι κάνουν και πώς φορολογούνται οι επιχειρήσεις οι ειδικές και οι κινέζικες και πώς φορολογούνται οι δικές μας ε, δεν θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί Γι' αυτό να σκεφτούμε λίγο την φορολογία και να δούμε τι γίνεται και με τον τελικό πελάτη. Γιατί όλα τα προϊόντα όλου του πλανήτη έρχονται στην ε, ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο για να είναι και ανταγωνιστικοί και οι εργαζόμενοι. Μην φορολογούμε τον εργαζόμενο συνέχεια και την επιχείρηση. Ευχαριστώ η κυρία Τράουτμαν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό θα, δώσω, θα μεταφέρω στην Επιτροπή ένα πολιτικό μήνυμα μετά από την άριστη εργασία του συναδέλφου εδώ είναι ιστορική καμπή πολιτική γιατί δεν χρησιμοποιούσαν αυτό τον όρο της βαμβικής πολιτικής ε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμα κάτι δεύτερο. Η στρατηγική του 2020 δεν επήρε στα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όλα αυτά τα σχέδια που ανακοινώθηκαν δεν δημιούργησαν και πολλές ελπίδες ε, εδώ για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας θα πρέπει να επηρεάσουμε την απασχόληση. Δεύτερο, να δούμε μια, μια κάθετη πολιτική που θα καλύπτει τα πάντα και όχι μόνο με τις δραστηριότητες διαφόρων τομέων, αλλά να έχουμε να κάνουμε με κάθε τομέα και με κάθε τομέα που αφορά και την Επιτροπή, όπως και τις δημόσιες αγορές και τον ανταγωνισμό. Χρειάζεται συνοχή από πλευράς Επιτροπή να δειχτεί για ένα πολιτικό συντονισμό των κρατών μελών μα. Κάτι ακόμα να επιμείνω σε τομεί κλειδιά. Αν επιθυμούμε οικονομική πολιτική που ε, καλή. Θα πρέπει να δούμε, να προσέξουμε τις τομείς που αλλάζουν όπως την αυτοκινητοβιομηχανία, ε, τα φάρμακα, που τις καινούριες άδειε για καινούρια μοριακά φάρμακα και επίσης ιδιαίτερα να προσέξουμε τις μεταφορές, τις τρομικές μεταφορές, ε, την πράσινη τεχνολογία και επίσης την ψηφιακή τεχνολογία και όλο τον τομέα των τελεπικοινωνιών Αυτή είναι από τους τομείς κλειδιά που θα πρέπει κύριε Πρόεδρε να προκαλέσουμε ξεκινήσουν ε, μια συζήτηση για τα μέσα που διαθέτουμε. Με τα λεφτά που έχουμε μπορούμε να το κάνουμε, με τα κονδύλια αυτά. Όχι, χρειάζονται ειδικά ταμεία, ώστε στου τομεί αυτή να έχουμε, αυτούς, να έχουμε δυνατότητα οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να μπορούν να έχουν τα μέσα για να αναπτύξουν και τι άλλε εκμεταλλευσή του με τι γνώσει του, με την παραγωγή του τη σωστή. Εδώ αυτή η κρίση κάτι δείχνει απλά και μόνο ότι δεν θα ξεφύγουμε από αυτή μόνο με μια εξυγίαση δημοσιονομική. Χρειάζεται να πουλήσουμε και προϊόντα και όταν βλέπουμε άλλες ανταγωνιστικές χώρες ε, να οργανώνουν την αγορά τους ε, και συστήματα ε, κατάλληλα πλαίσια και να μην μπορούμε εμεί να παρέμβουμε από τη στιγμή που είμαστε ανταγωνιστικοί δεν πρέπει να είμαστε αφελείς χρειάζεται να είμαστε περισσότερο οργανωμένοι σε σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων, τα ευρωπαϊκά όπως επίσης και των επιχειρήσεων παντού για να είμαστε περισσότερο αξιόπιστοι επίσης απέναντι στους πολίτες Ευχαριστώ. Ο ε, χρόνος πιέζει, τελειώνει η συζήτηση εδώ πέρα. Ε, λυπούμε, δεν γίνεται αλλιώ. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Η συνάδελφος δέχτηκε να αλλάξει και η σειρά τη ημερήσια διάταξη. οπότε νομίζω πρέπει τα επόμενα 20 λεπτά να τα αφιερώσουμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη ε, να με συγχωρείτε, δεν γίνεται αλλιώ. Ακούσαμε τον κύριο Λάγκε, τώρα θα τα υπόλοιπα θα τα δείτε με τους συντονιστές. Ε, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Λοιπόν, η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα έχει τον λόγο και έχουμε 20 λεπτά όπως σας είπα να περιοριστείτε όλοι σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ομολογώ ότι είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη μια που χθε έλαβα ένα τηλεφώνημα με πήρε τηλέφωνο η γραμματεία και μου είπαν να αναβάλω την παρουσιασή μου γιατί ο κ. Λάγκε πρόκειται να αποχωρήσει. Επαναλαμβάνει να αλλάξω την ημερομηνία γιατί ο κύριος Λάγκε ε, ε, επρόκειτο να σπεύσει να αναχωρήσει και ε, πρέπει να πάρω πρώτη τον λόγο και επίσης μου υπεσχέθησαν ότι η συζήτηση για το κείμενό μου επρόκειτο να κρατήσει μία ώρα τώρα προκύπτουν άλλα μόλις ένα το τώρα μου απομένει για να το ξεκαθαρίζουμε ευθύ εξ αρχή, είπαμε λίγο πρώτα θα έχουμε για κάθε σημείο μία ώρα. Ε, πάρα πολύ καλό το ότι μα τα είπατε και τώρα το αλλάξαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα δε έχουμε το, ένα άλλο πρόβλημα ότι πάρα έχουμε χρόνο από πέρυσι. Τέλο πάντων. 20 λεπτά, ε, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτά τα 20 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως ε, που μας δώσετε δυνατότητα να κάνουμε την ε, αλλαγή. Νομίζω χρειάζεται ο χρόνο. Do you hear me now? Τώρα ακούγαμε. Για να σας τα πω στα αγγλικά. Πρώτα πρώτα, να ευχαριστήσω Πρόεδρε, άπαντες, όλους μας τους συνεργάτες όλους που με βοήθησαν να συντάξω την έκθεση. Τη γραμματεία, του συμβούλους μου, του, του συνεργάτες μου, επίσης ευχαριστήσω την Κομισιόν και τον ε, ε Γενικό Διευθυντή, διότι συνεργαστήκαμε, έκαναμε ένα σωρό συναντήσεις για το θέμα μας και επίσης να ευχαριστήσω τους κοιόδης ηγητές ε, και όλους ε, από εσάς που έχετε στείλει, κάποιες ε, παρατηρήσεις. Με τις δίκες της Αβώνας τώρα ξεκινάει μια καινούργια περίοδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε η ώρα να προσαρμόσουμε ε, τους στόχους μας και τις προτεραιότητες μας ε, με τη συνθήκη. Σήμερα συζητούμε την ε, στατική αυτή όπως την έχει γονίσει η Ευρωπαϊκή που είναι η πρώτη μετά την ε, συνθήκη για να δούμε πώς θα υλοποιηθεί το άρθρο 194. Δηλαδή, αυτή η οριστική ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να διέπεται από υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και κανένα κράτος μέλος να μην αναγκαστεί να χάσει το τρένο. Και αυτή η στατική που εξεπώνησε η Κομισιόν πρόκειται να ενδυναμώσει, να αναβαθμίσει την πολιτική μας ως εξή. Πρώτον, τώρα θα ολοκληρώσουμε την ενεργειακή αγορά. Δεύτερον, θα έχουμε εξυγχρονισμό των δικτύων και της υποδομής. Τρίτον, οι δυνατότητες μας για αποτελεσματικότητα ενεργειακή πρόκειται να αποδώσουν. Θα πρέπει πάντως να έχουμε ένα στενό σύνδεσμο και συνεργεία μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ενεργειακής πολιτικής. Η δε ασφάλεια που απαιτείται ε, προϋποθέτει αυτήν την σχέση. Έρευνα και καινοτομία επίσης να προσέξουμε για να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά την εσωτερική αγορά και την ολοκλήρωσή της ευρωπαϊκή πολιτική. Μας έχει τονίσει ότι χρειάζεται επιγόντω να εφαρμοστεί το κοινοτικό δίκαιο και έχει δίκαιο και το δεύτερο ενεργειακό πακέτο και πρέπει να δούμε πώς θα πάμε και στην εφαρμογή του τρίτου πακέτου. Όμω δεν πάνε καλά τα πράγματα και γι' αυτό θα πρέπει να έχει πάρα πολύ αυστηρή στάση Κομισιόν για όσου κυβερνήτε δεν κάνουν και πολλά πάνω σε αυτό. Επίση να δούμε πώ η οδηγία θα γίνει κανονισμό. Αυτό ήδη έχει συμβεί στο παρελθόν. Και επίση έτσι θα πρέπει να δούμε πώ θα γίνει η δεύτερη έρευνα της Κομισιόν για τον κλάδο. Να δούμε Πώς θα αποδώσει η νομοθεσία, γιατί και οι καταναλωτέ και οι επιχειρήσεις θέλουν ένα σταθερό περιβάλλον ακριβώς λόγω της τάξης μεγέθους των χρημάτων που έχουν επενδυθεί σε έργα ενεργειακά. Όμως, επίσης θα πρέπει κάτι να κάνουμε όσον αφορά το, τις συνέπειες, μη εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές και ξεκαθαρίζω στον γραφό της Κομισιόν ότι η εσωτερική αγορά δεν θα λειτουργήσει σωστά χωρίς μαζικές επενδύσεις στις επενδύσεις και στα δίκτυα. Αν δεν έχουμε σύγχρονα δίκτυα, τότε υπονομεύεται το έργο μας. Τα έργα στο μέλλον θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο. Θα πρέπει η απαρχαιωμένη υποδομή να αντικατασταθεί ιδίω στις λιγότερο εμπτυγμένες περιοχές. Δύο είναι τα προβλήματα λέει Το ένα πρόβλημα είναι το δημοσιονομικό, το άλλο είναι το διοικητικό. Από πλευρά διοικητική είναι σαφέ ότι το ΤΕΝ δεν μα καλύπτει. Άρα θα πρέπει να αντικατασταθεί, όχι απλώ να αναθεωρηθεί. Χρειαζόμαστε σε κάθαρε προτεραιότητε κυρίως για την ε, επιλογή έργων και προγραμμάτων. Για να δούμε τι θα κάνει η Κομισιόν. Και θα πρέπει να έχουμε και κάποιες ε, προτάσεις, να τις μελετήσουμε, αυτές που διατυπώνω στην εκθεσή μου. Το δημοσιονομικό είναι ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα, ιδίω στον κλάδο της ενέργειας. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αυστηρό ο προπολογισμό, ότι υπάρχει σπάνιση στου πόρου. Όμω πρέπει να έχουμε ξεκάθαρου πολιτικού στόχου και αντίστοιχε αποφασιστικέ ενέργειες και αποφάσεις. Αυτό αποτυπώνεται στις ε, προοπτικές, στις μισομικές, αλλά θα πρέπει να δούμε πού αλλού μπορούμε να βρούμε τρόπους ε, χρηματοδότησης αυτών των μεγάλων επενδύσεων, όπως ας πούμε εγγύησει δανείων. Ας πούμε έχουμε τον, τον ΠΕΠ ε, τους κανόνες που μας οδηγούν σε ένα πρόγραμμα ενεργειακό μεγάλο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για, το, για τη σύνθεση του ενεργειακού τους πακέτου, το Energy Mix. Εν ώψη της πολιτικής 2020 πάντως θα πρέπει να έχουμε και περισσότερη έρευνα για, ε, για βιομάζα, για, για φυσικό αέριο, για εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. και το αέριο από πετρώματα θα πρέπει να μελετηθεί και να δούμε ε, για αυτό το αέριο από πετρώματα πώς μπορούμε να έχουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα. Ήρθε η ώρα να υλοποιήσουμε την απόφαση του 2008 τόσο ώστε να δημιουργήσουμε μια ανανεώσιμη αγορά πανευρωπαϊκή για την ενέργεια. Και γιατί επιμένουμε στο Βορρά όπου εκεί έχουν περιορισμούς λόγω κλίματος, λόγω γεωγραφίας και όχι και στο νότο όπου η μέρα είναι πιο μεγάλη, έχει περισσότερο ήλιο Να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε και το, το άνεμο, το αιωλικό στοιχείο και ο τόπος η των ενεργοστασίων να μην καροθορίζεται από τα σύνορα αλλά με το που θα είναι πιο αποδετικά. Και να δούμε πώς θα διευκολύνουμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι άλλο που τονίζει η Κομισιόν είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν το θίγω για μακρόν στην έκθεση γιατί έχει γίνει στην έκθεσή μας μια έκθεση για το θέμα. Ελπίζω πάντως ότι η Κομισιόν τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής θα λάβει υπόψη αυτά που μας λέει εδώ. Για την αποτελεσματικότητα έχω να πω ότι χρειάζεται μια κοινή μεθοδολογία πριν πάμε σε δεσμευτικούς στόχους. Και να έχουμε δεσμευτικούς στόχους μόλις αποφασίσουμε το πώς θα μετρούμε, πώς θα ελέγχουμε τους εθνικούς στόχους. Για την ε, ασφάλεια ενέργειας θα πρέπει να ζητήσουμε κάποια διαφάνεια από τους ε, εταίρους μας. Και αυτό είναι βασικό σημείο τη έκθεση διότι είναι σαφές πως συνδέονται εσωτερική και εξωτερική ενεργική πολιτική. Έχουμε αέριο και πετρέλαιο που το εισάγουμε. Γι' αυτό και θέλω οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς να επεκταθούν όσο γίνεται περισσότερο σε σχέση με τους ε, εταίρους μας από το εξωτερικό. Οι ξένες εταιρείε που έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να βρίσκουν περιβάλλον ρυθμισμένο και με διαφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για τους αγωγούς που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και εκεί θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχους κανόνες που να διέπουν την ύπαρξη τη λειτουργία τους κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Ο Επίτροπος καιρό όταν απάντησε σε μια έγγραφη ερώτηση που είχε υποβάλει ε, και είπε προς τον το τύπο ότι έτσι βλέπω τα πράγματα, έχει τις ίδιες απόψεις. Όμως, σας τονίζω ότι αυτή η διαφάνεια θα πρέπει να αφορά όλους τους αγωγούς, όλους σημερινούς, αυριανούς και όχι ορισμένους εξ αυτών. Σας τονίζω ότι χρειάζεται μια μακρόπνοη πολιτική. Ένα όραμα μακρόπνο, ώστε να φτάσουμε όσο γίνεται σε περισσότερο ενιαία ε, ενεργειακή πολιτική και να υπάρχει υπευθυνότητα, να υπάρχει αλληλεγγύη. Ο κ. Μπούτζεκ το λέει αυτό μια νέα ενεργειακή κοινότητα, άλλοι το λένε το, το ΝΑΤΟ της ενέργειας, Όπω θέλετε να το ονομάσετε. Όπως Όμως, όσο νωρίτερα το καταφέρουμε, τόσο καλύτερα. Αυτή η δεκαετή στρατηγική νομίζω θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Uh, ε, δώσα μένα get δώσαμε να δώσω το λόγο. Ε, ε, Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μπομπίνσκα για, για το έργο της και βεβαίω ζητάμε και συνεισφορά από άλλε ομάδες λοιπόν ως σχεδισηγήτρια των σοσιαλιστών θα ήθελα να πω πως η έκθεση αυτή έχει πάρα πολλά θετικά σημεία συμφωνώ πως ε, Οπωσδήποτε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπληρώνουν ε, τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτό είναι σημαντικό για να επιτύχει η πολιτική αυτή. και βεβαίως ε, για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα πράγματι σωστό είναι πως ε, υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σχετίζεται και με τα νοικοκυριά και με τους πόρους ε, και υπάρχει πολιτική συμφωνία 100% πως είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα αλλά ταυτόχρονα λίγα πράγματα γίνονται οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως τόνισε η συγκήτρια να υπάρξει αποτελεσματική χρήση των πόρων. Εγώ θα ήθελα να δω βελτιάσεις, βελτιώσεις στο κομμάτι κλίματος, αηφορίας και καταναλωτών. Εκεί θα κάνω κάποιες ε, τροπολογίες για την πολιτική του κλίματος, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πρέπει να τονιστεί, αναφέρεται στην έκθεση αλλά η ισορροπία διαταράσσεται από τις ε, παραδοσιακές ε, πηγές ενέργειας ε, που βλέπουμε εδώ πέρα το αέριο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αλλά οι ανανεώσιμες πρέπει να τονιστούν γιατί πρέπει να είναι σαφές πως η ενεργειακή στρατηγική πρέπει να, να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την κλιματική πολιτική. Αυτό είναι σημαντικό και για τη βιομηχανική πολιτική που αναφέραμε πριν, για την ε, αντιαγωνιστικότητά μας στο μέλλον και η ενεργειακή στρατηγική μας επιτρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 25 έως 30% και θα κάνω εγώ τις αναλογίες τροπολογίες και θα πρέπει να δούμε μια τιμή για το διοξίδιο του άνθρακα που θα αντισταθμίζει αρνητικές ε, εξέλιξεις και εκεί πέρα πρέπει να δούμε την οδηγία για τη φορολογική ενέργειας Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση ε, το κομμάτι για τους καταναλωτές. Δεν αναφέρονται αρκετά. Γνωρίζουμε πως υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού και άρα οι είναι πολύ ψηλές πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια γιατί είναι πολύ ψηλέ τιμέ. Ε, Όπω είπε λοιπόν και η συνάδελφο, πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα του καταναλωτή. Πρέπει να γίνει λοιπόν πιο σαφέ εδώ πέρα και, και τι. Αυτό να αφορά και τα προϊόντα τα χρηματοπιστωτικά. Βεβαίω αυτό είναι άλλο θέμα από αυτό το οποίο συζητάμε. Πρέπει λοιπόν να χτυπήσουμε και τα μονοπόλια. Οπότε προ τα εκεί θα πάνε οι παρεμβάσει μου. Και ένα τελευταίο κομμάτι από μένα. Τελευταία παρατήρηση. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη σαφού ε, δήλωση για τι επενδύσει, αλλά μπορεί να ενισχυθεί ακόμα παραπάνω. Σύμφωνα με τα όσα είπε η συγκήτρια. Και χρειάζονται Βεβαίω επενδύσει στι υποδομές γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους άλλους τομεί αυτή τη πολιτική. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει κάποια κονδύλια. Για να ενισχύσουμε σε αυτά τα οποία λέει η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για το έργο της και για την ε, ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στη διαδρομή αυτή. Είναι πολύ καλό το σχέδιο και συμφωνώ σε επιτοπλίστων με την έμφαση που δίνεται στην ε, εφαρμογή της ισχύουσης νομοθεσίας και των σχετικών πρωτοβουλειών ή στην εσωτερική αγορά και όσον αφορά την εξασφάλιση της ε, ενέργειας. Όπως λέτε και σωστά θα πρέπει να είμαστε όμως και έχουμε μια τροπολογία όπου προσθέτουμε κάποιες ε, ε, απόψεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση, κάποιες πράσινες μόρφες ενέργειας, ανανεώσιμες, ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και όλες αυτές οι ιδέες νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να τις αναπτύξει περισσότερο, όμως πάντως καταρχήν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιολόγο το σχέδιο κειμένου και περιμένουμε καλή συνέχεια. Και εγώ θα πρέπει να είμαι σύντομο. Ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή. Θα πρέπει να έχουμε κάποιες ε, προσθήκες. Θα ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τα θέματα του ανταγωνισμού στην παράγραφο 8. Τι γίνεται δηλαδή σε σχέση και ποια είναι η σχέση των συναρμοδίων αρχών ανταγωνισμού με τις κανονιστικές αρχές. Επίσης, μπορώ να συμφωνήσω για το ότι αυτοί που κάνουν τις μεταφορές της ενέργειας είναι πολλές φορές κρατικοί φορείς. Δηλαδή θα πρέπει να καλυφθούν και αυτοί. Και αυτοί οι φορείς, οι κρατικοί. Προσέξτε, οι Ιταλικές εταιρείες λένε για 5.000 μεγαβάτ το οποίο σε Μαυροβούνιο, την Ισία, Αλβανία παράγεται από αυτούς και επανεισάγεται μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι συμβαστό με, το, με την πολιτική μας. Θα πρέπει επομένω με το σύστημα που έχουμε Θα πρέπει να συνδέσουμε όλους αυτούς τους τόπους μέσα πρωτοβουλίε παρουσμετοίτιες e και κάπως να ρυθμίσουμε το θέμα των εισαγών ενέργεια. Όσον αφορά τώρα την εξασφάλιση προμήθεια ενέργειας, προσέξτε το εξή. Η εξάρτηση μας μεγαλύτερη είναι σε σχέση με το πετρέλαιο και σε σχέση με την Ρωσία. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εισάγουν πάρα πολύ δίζελ ψηλής ποιότητας από τη Ρωσία. Επομένω, θα πρέπει κανείς εκεί να προσέξει, εκεί να φοβάται τι γίνεται με την εξάρτηση. Φτάνουμε μέχρι το 89% για κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Άλλα δύο θέματα που δεν μου άρεσαν τόσο πολύ. Παράγραφος 26 όσον αφορά την αποτελεσματική σχέση της, στη χρήση της ενέργειας το 2003. Είχαμε πει ότι πρέπει να κοινή μεθοδολογία. Αλλιώς δεν θα έχουμε ε, ε, στόχους δεσμευτικούς. Το 2003 λοιπόν είχε γίνει αυτή η οδηγία για ενέργεια και, ε, και υπηρεσίες. Κοινή μεθοδολογία θέλει η Κομισιόν. Όμως τα κράτη-μέλη είπαν όχι στις διαπραγματεύσεις. Μετά είπαμε να αρχίσει μια επιτροπολογία. Η Κομισιόν πρότεινε μια κοινή μεθοδολογία. Κάποιοι κρατημέλοι όμω ε, άσκησαν βέτο κατά την επιτροπολογία και βρισκόμαστε τώρα πέντε χρόνια μετά από αυτήν την οδηγία για τις υπηρεσίες να έχουμε αυτό το βέτο των κρατών μελών. Αν δεν υπάρχει κοινή μεθοδολογία μπορούν να κλέβουν τα κρατη να κάνουν ζαβολία στο σύστημα. Και σε πολλές χώρες το 50% αυτά το οποίο ζητούμε σήμερα το έχουν κάνει από δεκαετία του 90. Αν λοιπόν εμείς σε κάποια παράγραφο του ψηφίσματος της εκθέσεως να πούμε στις κυβερνήσεις ότι αν δεν υπάρχει μεθολογία, δεν υπάρχουν και δεσμευτικοί στόχοι. Και έτσι κάτι θα κάνουμε για αυτή τη σκανδαλώδη πολιτική κάποιων κρατών μελών. Αλλιώ εξαρτώμεθα από, από το αν θα πετύχουν ή όχι τα κράτη-μέλη. Τώρα το άλλο είναι για το κατά πόσο θα έχουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με χρήση πανευρωπαϊκή. Κοιτάξτε εγώ, επί 1,5 χρόνο μεταξύ 2008 και τέλος του 2009 πέρασε όλη αυτή την περίοδο κουβεντιάζοντα αυτό το θέμα και καταλήξαμε ότι σήμερα τα εθνικά συστήματα υποστήριξης είναι καλύτερα και μακροοικονομικά από οποιοδήποτε άλλο σύστημα πιστοποίησης. και άλλωστε στην οδηγία προβλέπεται αναθεώρηση του 2014 και θα αναλυθεί ξανά το θέμα. Οπότε ίσως είναι κάπως ε, πρόημο. Θα έχουμε το 2010 στην εθνικό επίπεδο ε, εφαρμογή της οδηγίας. Επομένως, γιατί να ξανανοίξουμε αυτό το θέμα το τόσο δύσκολο, το πόσο περίπλοκο και να δημιουργήσουμε στους επενδυτές μία ανασφάλεια. Γιατί όταν έρθει η ώρα χρειάζονται πιστώσει από τι τράπεζε και επομένω θα πρέπει να, είναι ευδιάκριτα, προβεβλημένα τα συστήματα υποστήριξη. Αυτά είχα να σα πω σαν ιστορικό πλαίσιο για το θέμα μα. Ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση υπόσχεται πολλά και μας αρέσει το ότι σε αυτή την έκθεση εστιάζεστε στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Έχουμε μονοπόλιο στην αγορά. Έχουμε συρρήκνωση του ανταγωνισμού. Έχουμε αυτές τις επανεξαγωγές, χρειάζεται μια ρήτρα ή επίσης απαγόρευση πρόσβασης τρίτων χωρών στην υποδομή του φυσικού αερίου. Και δεν έχουμε θέμα μόνο φυσικό έχουμε και θέμα άνθρακα που έχει ακόμα σημαντικό ρόλο στην ισορροπία των ενεργειακών πόρων. Τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια όλοι μας λένε πρέπει να εγκαταλείψουμε τον άνθρακα. Αυτό είναι κατανοητό, αν λάβουμε υπόψη την ενεργειακή πολιτική, αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε κόστος. Δεν θα πρέπει να γίνει με το να ευνοούμε περισσότερο τα μονοπόλια και περισσότερο την εξαρτησή μας. Άρα πρώτα να κάνουμε μια μεγαλύτερη κατάδυμη των αναγκών μας και μετά. Αυτό ισχύει για και την Ανατολική Ευρώπη. Αλλιώς θα είναι μεγάλο λάθος να προχωρήσουμε με άλλο τρόπο. Αυτό τονίζεται στην έκθεση. Ευχαριστώ. Έχω πέντε ακόμα ομιλητές και ο Γενικός Διευθυντής ήρθε και περιμένουν οι Υπουργοί. Η κυρία Ποδηματά μου λέει μήπως ε, μπορούμε στην επόμενη συνεδρίαση όσοι είναι τώρα στον κατάλογο να μιλήσουν πρώτοι στην επόμενη συζήτηση. Ίσως να κάνουμε αυτό. Αλλά ίσω να ακούσουμε πρώτα απ' όλο τον κύριο Γενικό Διευθυντή. Αλλά και η κυρία Ποδηματά θέλει να πει κάτι επί τη διαδικασία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Επειδή συμμερίζομαι απολύτω αυτό που είπε η συγγήτρια καταρχήν, για αυτή τη συζήτηση θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον μία ώρα στη διάθεσή μα. Και επειδή είναι σημαντικό να μπορέσει το κοινοβούλιο αξιοποιώντας και το νέο θεσμικό του ρόλο στο πλαίσιο της συνθήκης να επηρεάσει τις συζητήσεις που γίνονται στο συμβούλιο αυτή την περίοδο για το σχεδιασμό της νέας ε, ενεργειακής στρατηγικής της ευρωπαϊκής ένωσης. γι' αυτό το λόγο λοιπόν προτείνω εκτάκτως να διασφαλίσουμε μισή ώρα στην επόμενη, σύνοδο της επιτροπής μας 29 και 30 σεπτεμβρίου για να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο αυτή η εξαιρετικά σημαντική συζήτηση. Ωραία, θα το δούμε με τους συντονιστές. Έξυπνη πρόταση. Λοιπόν, ο κύριος Γενικός Διευθυντής, έχετε τον λόγο και με συγχωρείτε που έχετε τόσο λίγο χρόνο. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή σας και την εισηγήτρια. Αυτό το κείμενο που το επεξεργάζεται νομίζουμε θα συμβάλλει πάρα πολύ όσον αφορά τις επιλογές που έχουμε για να χαράξουμε την πολιτική που θα υποβάλουμε τον Νοέμβρη και θα έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την επόμενη δεκαετία για το ενεργειακό βεβαίω και θα επανέλθουμε όποτε θέλετε για να τα ξαναπούμε προετοιμάζοντας αυτό το ψήφισμα τώρα να μην επαναλάβω όσα φύγει η, έκθεση, τα θέματα τα οποία πάντοτε συμφωνούμε εσείς και εμείς ε, ιδίως όσον την εφαρμογή της ελληνικής αγοράς, τις επενδύσεις για τα δίκτυα. Όμως, πέραν αυτού, ο εξυγχρονισμός των υποδομών είναι πάρα πολύ βασικός, ούτως ώστε να μπορέσουμε τις ενωμένες πηγές ενέργειας να τις βάλουμε και να τις εντάξουμε στο σύστημα και χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν σε παγκόσμια κλίμακα για να μειώσουμε τις πηγές ενέργειας. Και έτσι θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις ανάγκες μας, όπως είπε ο κ. Σιμάνσκι και την εξάρτησή μας. Περιμένουμε να ακούσουμε από το Κοινοβούλιο τι λέτε για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και να δούμε πόσο πιστεύετε χρειάζονται δεσμευτικοί στόχοι για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Ακούσαμε την συγκίτρια για το ότι έλαβε υπόψη τους καταναλωτές στις δικές ε, αγορές και το ότι χρειάζεται μια συνολική άποψη της ενεργειακής πολιτικής στα πλαίσια των ε, πολιτικών που προτείνουμε. αλλά και κλίματος, ενέργεια, φορολογική πολιτική. Άρα με την κυρία Χίντεγκαρτ θα προχωρήσουμε σε στενή συνεργασία και με τους άλλους αναμόδους αδέλφους και όποτε νομίζετε να ξανάρθουμε για να ξεκαθαρίσουμε και άλλα θέματα, γιατί έχουμε εδώ κάποιες τεχνικές προτάσεις. Ε, έχουμε αυτές τις προτάσεις που αφορούν ε, το φυσικό αέριο, που αφορούν τον άνθρακα. Αυτές τις προτάσεις μπορεί να υποβληθούν γράφους αν θέλετε. Σας ευχαριστώ για το ότι θα μας τα στείλετε και γραπτός και υπενθυμίζω πως η προθεσμοί για τις τροπολογίες είναι η 7η Σεπτεμβρίου και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια ε, και συγγνώμη. Ε, έχετε δίκιο πράγματι. Πρέπει όλοι να είμαστε κάπως πιο πειθαρχημένοι έτσι ώστε αυτοί που είναι τελευταίοι στη μερίσια διάταξη να μην ε, είναι συνεχώς αδικημένη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Η Βέλγια Υπουργή είναι εδώ και παρακαλώ λοιπόν να περάσουμε αμέσως να προχωρήσουμε παρακάτω στο μερίς και διάταξη. Κυρίες ε, και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Καθίστε για να ξεκινήσουμε. Ζητώ συγγνώμη από τους υπουργούς γιατί περίμεναν. Λοιπόν, τώρα θα μαζέψουμε μαζί τις ερωτήσεις για να κερδίσουμε το χρόνο. Καλώς ορίζω την κυρία Ζαμπίν Λάριουελ, Υπουργού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Αυτοαπασχολούμενων Γεωργίας και Πολιτικής Επιστημών και τον Φίντσεντ Φαν Κβίκενμπορν, Υπουργό Επιχειρήσεων και Απλοποίησης. Λοιπόν, θα κάνουν κάποιες σύντομες δηλώσεις οι Υπουργοί και μετά θα συζητήσουμε. Θα ξεκινήσει η κυρία. Βεβαίω η κυρία θα ξεκινήσει. Ναι, θέλουμε, θέλαμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με πραγματικά προγράμματα αποτελεσματικά που να είναι υπέρ του πολίτη και να συνεισφέρουμε στους στόχους, στην επιτυχία τους όσον αφορά την κοινοτομία και την έρευνα. Το οικονομικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι δύσκολο και μάλιστα σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι οι έρευνες σε αυτό συγκεκριμενοποιούνται πάντα μέσω βελτιώσεων στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Στη στρατηγική του 2020 αυτή η πολιτική για τον ζωτικό αυτό χώρο μπορεί να βοηθήσει για την ανάπτυξη, για την βελτίωση των πραγμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει αποδειχθεί ότι θα μπορούσε να προσφέρει ο τομέας αυτό αυτός σημαντικά εργαλεία για την πρόκληση την παγκόσμια όπως για την αλλαγή του κλίματος, για την ανάπτυξη. Το 189 άρθρο κύριε Πρόεδρε και δεν είναι κάτι το καινούριο που σας λέω προβλέπει νέο, νέα εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει πώς θα συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Ινστιτούτο και η μελλοντική ανάπτυξη αυτού βέβαια θα αποτελέσει αντικείμενο σύνταξης έκθεσης από την Επιτροπή της 20 Οκτωβρίου και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι μια σημαντική πτυχή και σταθμός στην πολιτική αυτή την ευρωπαϊκή. Εμείς θα προσέξουμε τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα, κάτι το σημαντικό κατά την απόψή μου, είναι να προχωρήσουμε για μια ευρωπαϊκή ενόραση για την εκπλάση του διαστημικού χώρου ακριβώς χάρη στις Ευρωπαίους εταίρους. Για να δούμε από τεχνολογικής πλευράς τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα γίνει και με τα απαραίτητα κονδύλια για αυτό το φιλόδοξο κοινό μας στόχο. Πώς αυτή τη νέα εταιρική σχέση σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορέσουμε να την οργανώσουμε. Πολλά τα θέματα αυτό σε μια συνάντηση 21 Οκτωβρίου σε υπουργικό επίπεδο στο Μέγαρο Egmont. Θα οργανωθεί αυτό και θα δούμε και από τεχνικής πλευράς ε, την οργάνωση και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και ταυτόχρονα θα θέλαμε και τη δική σας βοήθεια από την Επιτροπή σας. Ε, σίγουρα βέβαια ε, είστε και προσκεκλημένοι σε αυτή τη συνάντηση μετά στην στην διαρκή χρήση Γαλιλαίου και GMS και με το πρόγραμμα αυτό που δείχνει πώς αυτές οι διαστημικές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τον Ευρωπαίο πολίτη και ιδιαίτερα τα προσέχουμε αυτά και θα τα προσέξουμε τις έξι μήνες προεδρίας μας και οι προκλήσεις είναι κυρίως οικονομικές, τα κονδύλια για το με αυτό. Τρίτο, η διαστημική πολιτική είναι ενταχθεί στην πολιτική ασφάλειας και με όσα έχουν να κάνουν βέβαια και με τις κλιματικές αλλαγές. Κάτι τέταρτο, ιδιαίτερα σημαντικό, εμείς ε, θα θέλαμε να ενισχύσουμε το ρόλο αυτό των διαστημικών εργαλείων στη στρατηγική ε, φύσεως συνεργασία με την Αφρική και τηλεπικοινωνίες, παρατήρηση της γίνης επιφάνειας, τηλεπικοινωνίες, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Αφρική και θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικών εφαρμογών για την Αφρική πολλές πρωτοβουλίες ε, και των Αφρικανών εταίρων θα υποστηριχτούν από εμά. Όπως και για την πολιτική ανάπτυξη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που ε, προσφέρουν αυτά τα διαστημικά προγράμματα. Είναι λοιπόν σημαντικό για την Αφρική και στις 16 Σεπτεμβρίου οργανώνεται σε ανώτερο επίπεδο μία συνάντηση με την ΕΖΑ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους ε, Αφρικανός εταίρος για την ε, καινοτομία, την τεχνολογία κλπ. 20 Σεπτεμβρίου το Space Council θα χαράξει τους προσανατολισμούς ε, σε αυτές, ε, προς αυτήν την κατεύθυνση. Τον καλέο και τον Τζίμες θα δούμε την αναπτυξή τους όπως επίσης και τα θέματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και για την ασφάλεια του διαστήματος που είναι μια πραγματική για μας πρόκληση με τη ισχύ της ε, συνθήκη της Αβώνας και με την ανάπτυξη αυτή, την εξέλιξη, την οικονομική του δεύτερου μήνες, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Θα πρέπει να δούμε σε διαστημικό επίπεδο, σε παρόμοια θέματα, πώς θα υποφεληθούμε από κάθε ευκαιρία. Η θέση απέναντι στην ΕΣΕ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και θα μπορέσουμε να, ε, να αποτελέσει το διάστημα γίνεται πιο ψηλά μεταφορικά και πραγματικά στο χρονοδιάγραμμά μας και να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά τα διαστημικά. Και η ΕΖΕ βέβαια έχει διαθέτει ιδιαίτερη πείρα και ρεαλιστική αντιμετώπιση που τη χαρακτηρίζει και θα πρέπει να διαχειριστούμε το διαστημικό χώρο μέσω της πύρας και των επενδύσεων στα χώρες μέλη του ΕΣΑ και τα κράτη-μέλη αυτά θα πρέπει να προσκληθούν να συνεχίσουν τη χρηματοδότησή τους όλων αυτών των εργαλείων. Με λίγα λόγια κύριε Πρόεδρε, αυτές ήταν τέσσερις μεγάλες ιδιαίτερε προτεραιότητες, βασικές προτεραιότητες από δικής μας πλευράς Βελγίου για το διαστημικό χώρο. Ευχαριστώ. Πράγματι θέσατε κάποια σαφή ζητήματα. Τώρα έχετε εσείς τον λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριοι βουλευτές. Εγώ θα σταθώ λίγο στις προτεραιότητες του Βελγίου στον τομέα των ε, τηλεπικοινωνιών. Γνωρίζετε πως ε, ε, βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή αφήνουμε πίσω μας ε, την ύφεση και βλέπουμε μεγάλο ανταγωνισμό από τις νέες αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό σημαίνει πως πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα η Ευρώπη και αυτό θα γίνει φροντίζοντας ε, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η ε, η οικονομία και βέβαια αυτό οι πληροφορίε ε, τηλεπικοινωνιών και πληροφορική παίζουν σημαντικό ρόλο. Ξέρετε πως ε, και η κυρία Κρούς δεν είναι μόνο αντιπρόεδρος κομισιών αλλά και αφορά, έχει συναρμοδιότητα στα θέματα της ψυχικής ατζέντας οπότε αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα θέματα και βλέπουμε πως ε, η πρώτη σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ατζέντα 2020 είναι η ψηφιακή ε, ατζέντα και όπως σας είπα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό το οποίο σημαίνει μια καλή αρχή για τα πράγματα οπότε το σημαντικότερο για την Προεδρία μας είναι να προωθήσουμε την ψηφιακή αυτή ατζέντα το αυτό πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε επί Ισπανικής ε, Προεδρίας και τώρα θα αναφέρω κάποιες ε, προτεραιότητες ε, τις οποίες θα προωθήσουμε. Πρώτα απ' όλα γνωρίζετε πως η ψηφιακή ατζέντα έχει πολύ φιλοδοξούς στόχους που βασίζονται και στην έκθεση της Επιτροπής σας κύριε Πρόεδρε υπό την ηγεσία της κυρίας Τεκαστηγιοβέρα πως δηλαδή πρέπει να επιτύχουμε αυτό τον στόχο μας ε, μέχρι το 2013 όπου ξέρετε πως αυτό σημαίνει πως μέσα σε 30 χρόνια θα πρέπει να έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι τη δυνατότητα ευρυζωνικού ίντερνετ και μέχρι το 2020 πρέπει να έχουμε μια κάλυψη 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού με αυτό το οποίο λέμε πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ. Μιλάμε για 100 Mbps. Οπότε πρέπει τα κράτη να κάνουν πάρα πολλές ε, προσαρμογές. Η ΔΕ Κομισιόν θα εγκρίνει τις ερχόμενες ε, εβδομάδες ε, το πακέτο αυτό της ευρυζωνικότητας. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τη στρατηγική της ευρυζωνικότητας με την ανακοίνωση της Κομισιόν που λέει πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, είναι έτοιμα με τα εθνικά τους σχέδια αλλά να δουν και βεβαίω εδώ είναι το σημαντικότερο πρόβλημα όταν μιλάμε για την ευρυζωνικότητα τα κονδύλια και θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα κράτη-μέλη αλλά και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για την ανάπτυξη της Υπέθρου. Νομίζω η ανακοίνωση Κομισιόν το πρώτο βήμα δεύτερο. Η πολιτική του φάσματος, ε, η σημασία που δίνουμε στο, ε, στην ασύρματη ευρυζωνικότητα. Ξέρετε πως ε, αυτό, σε αυτό θα αφιερώσουμε στις 22 και είχαμε με συγχωρείτε, 22 και 23 Μαρτίου ε, την Σύνοδο Κορυφής για το φάσμα και αυτό το οποίο προέκυψε είναι πως πράγματι ε, θα πρέπει να διαχειριστούμε με αποτελεσματικό τρόπο το ε, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα της δέσμες συχνοτήτων και να υπάρξει ένας κάποιος εναρμονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση το τι κάνουμε με το ψηφιακό αυτό μέρισμα το λεγόμενο με το switch off το λεγόμενο το σβήσιμο, τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση και τι θα κάνουμε με τα συγνότητες που απελευθερώνονται και πρέπει λοιπόν να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προσφέρουν και υπηρεσίες και βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία αφενός βεβαίως μέσω των αναγκών της ραδιοτηλεόρασης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Το άλλο κομμάτι βεβαίως ε, του πακέτου αυτή αφορά την πρόσβαση νέας γενιάς όπως λέγεται ε, πράγμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και μας απασχόλησε στη συζήτηση για το πακέτο το τηλεπικοινωνιακό υπό την πτυχή των επενδύσεων και βεβαίως αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τις επενδύσεις θα πρέπει να μπορούν να μαζέψουν τα απαραίτητα λεφτά για να το κάνουν αυτό και βεβαίως να υπάρχει και ο επαρκής ανταγωνισμός. Νομίζω πως εδώ πέρα η κυρία Τολκμένη έδειξε πολύ σωστά θέματα και θα πρέπει ακριβώς να ισορροπήσουμε αυτά τα δύο σημεία και βεβαίως ε, τις ερχόμενες ε, εβδομάδες ε, θα τα συζητήσουμε αυτά. Ένα κομμάτι ακόμα στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής το οποίο απασχολεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορά την ε, πιθανή επέκταση της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας για την ευρυζωνικότητα. Ξέρετε πως υπάρχει τέτοιο για το, κάτι τέτοιο για το τηλέφωνο και αναμένουμε βεβαίως την ε, Κομισιόν η οποία θα μας ενημερώσει για τις ε, πιθανότητες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ένα άλλο κομμάτι βεβαίως ε, αφορά την ασφάλεια του διαδικτύου και την ε, σχετική υπηρεσία την ΕΝΙΣΑ και εκεί πέρα η Κομισιόν θα καταθέσει προτάσεις ε, για το πώς θα λειτουργήσει και θα εξυγχρονιστεί η ενίσα στην ε, ψηφιακή ατζέντα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά πράγματα για το CRT αυτό το οποίο λέμε μία ε, ομάδα ανταπόκρισης εκτάκτου ανάγκης για τα ζητήματα αυτά πληροφορικής κάτι το οποίο θα αποτελέσει ευθύνη της ΕΝΙΣΑ. Τρίτο σημείο, έρευνα και καινοτομία στον τομέα αυτών. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν τρεις σημαντικές διασκέψεις. Έχουμε ένα, μία τον Σεπτέμβριο, δεύτερον μία σύνοδο κορυφής με μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 18 Νοεμβρίου και βεβαίως έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως ξέρετε το πρώτο θεματικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι αφιερωμένο στην έρευνα και την καινοτομία. Τέταρτον, σχέδιο δράσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ξέρετε, από το 2008 μέχρι το 2015 εγκρίναμε στο Μάλμε τη σχετική πολιτική για τα έτη αυτά για να φτάσουμε σε αυτό το οποίο λέμε διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες μας να εξυπηρετούνται από μία ψηφιακή αγορά, αν θέλετε, για τις υπηρεσίες αυτές και να είναι συμβατές μεταξύ τους αυτές η υπηρεσία και ξέρετε 16-17 Δεκεμβρίου προγραμματίζουμε και την ανάλογη διάσκεψη στις ε, Βρυξέλλες. Ε, θα τελειώσω με δύο πράγματα. Έχουμε το ζητηματίσει ουδετερότητες του δικτύου. Ξέρετε πως ε, ε, η Google και η Verizon στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έκαναν μια πρόταση για την ουδετερότητα του δικτύου. Ευαίσθητο ζήτημα, γνωρίζουμε πως υπάρχει διαβούλευση με την Κομισιόν και τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε και σχετική σύνοδο κορυφής. Πρέπει να τονίσω πώς επί Βελγικής Προεδρία, για εμάς λοιπόν στη Βελγική Προεδρία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό νομίζω το να είναι ε, οι ταχύτητες ίδιες για όλα τα site του είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Και τέλος, κάτι ακόμα κύριε Πρόεδρε, ε, κάτι το οποίο η Επιτροπή σας είδε με τρόπο εξαιρετικό και αφορά το όλο ζήτημα της περιαγωγής λογαριασμοί σοκ που έρχονται στους ανθρώπους ε, και υπήρχε βεβαίως ε, και απόφαση του ΔΕΚ ε, που κατέδειξε πως ήταν σωστή η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βλέπουμε λοιπόν πως για τα γραπτά μηνύματα και για την φωνή το έχουμε επιτύχει. Υπάρχει μια σαφής μείωση των τιμών, αλλά υπάρχει βεβαίως τώρα το θέμα των δεδομένων του κινητού ίντερνετ. Ξέρετε πως ε, είχαμε την έκθεση αυτού του Ιουνίου που αποδεικνύει πως το κόστος ε, ε, για ένα Μεγαμπάιτ είναι 2,6 ευρώ και μιλάμε βεβαίως όταν μιλάμε για ένα GB αν μιλάμε για βίντεο, φωτογραφίες κτλ δεν είναι τίποτα το φοβερό και οπωσδήποτε ε, βλέπουμε πως ε, για ένα γίγαμπάιτ για να κατεβάσει κανείς στο εξωτερικό χρειάζεται 2.600 ευρώ δηλαδή στο εξωτερικό έτσι μέσα στη χώρα είναι 80 ευρώ και εκτός της χώρας είναι 2.600 αντικειμενικά λοιπόν βλέπετε πως δεν μπορεί να εξηγηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω πως το Κοινοβούλιο και ειδικά η Επιτροπή σας θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες με αυτοπεποίθηση για να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Αυτά και γνωρίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μαζί σας και στις ακροάσεις ε, και εγώ έχω συναντηθεί και είχα πολλές καλές επαφές με τους ειδικούς για τις λεπικοινωνίες στην Επιτροπή σας και από κοινού με την Επιτροπή νομίζω θα φροντίσουμε για τα σημαντικά αυτά βήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριος Λάμπερτς πρώτα απ' όλα. Je voudrais euh, intervenir sur un dossier que ni vous, Madame Laruelle, ni vous, Monsieur Van Quickenborn, n'avez abordé. Θα μπορέσει μάλλον η συνάδελφος να απαντήσει, ίσως όμως και ο κ. Υπουργό. Θα ήθελα να μιλήσω κάτι για κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά στο Βέλγιο, τον άμελο νεκρούν Μπεστήρ. Αυτό είναι το θέμα περί της πρόσφατης ανάπτυξης, τώρα το καλοκαίρι, κάτι το πολύ ε, ενδιαφέρον βλέπουμε ότι έχουμε τρεις φορές παραπάνω χρήματα εδώ μιλάμε δύο από 2,7 δισεκατομμύρια προς 7,2 δισεκατομμύρια και στις ΗΠΑ ε, με 25% βλέπουμε ότι αποφασίζουν να απορρίψουν ένα πρόγραμμα. Εντάξει, εδώ λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε ε, ότι όσοι να παρόμοιο πρόγραμμα πρώτα θα τους απολύαμε και μετά θα το ξαναβλέπαμε και δεν θα το συνεχίζαμε. Θα πρέπει να συνεχίζουμε κάθε δυνατότητα. Αυτό που έγινε το Συμβούλιο τι αποφάσισε χωρίς να το πει αλλά το αποφάσισε τελικά ενώ το πρώτο κεραμίδι δεν έχει μπει στη σκεπή σε ένα σχέδιο που βλέπουμε ότι δεν ελέγχουμε που δεν είναι το κόστος και την αύξησή του έτσι τι γίνεται κάθε επιλογή μελετήθηκε όχι μόνο εντάξει για την Πρόμπερ ε, από τη στιγμή που θα πρέπει να το καταπιούμε το χάπι, τι να κάνουμε. Αλλά άλλοι είχαν πει όχι ούτε ένα, ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και από τη στιγμή που είπαν ότι ξεκίνησε αυτό και συνέχισε το Συμβούλιο, θέλησε να βρει τα χρήματα. Άλλο είναι να πούμε θα βρούμε τα χρήματα και άλλο είναι να πούμε πού θα τα βρούμε τα χρήματα. Δεν είναι μικρό ποσά. Μιλάμε για εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ. Από 2,7 περνάμε στο 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και με συμμετοχή ακριβώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε το Συμβούλιο ε, που δεν απάντησε μέχρι τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει, από πού θα τα βγάλουμε αυτά τα χρήματα, από ποιο πρόγραμμα, από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο πάνω απ' όλα. Πού θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα, επαναλαμβάνω. Μην τρέφουμε αυτά πάτες. Ε, αυτό που θα το δώσουμε ε, παραπάνω εκεί θα το φέρσουμε από άλλα προγράμματα. Ναι, λοιπόν αυτό πολύ σημαντικό για να δούμε τι θα κάνουμε, ποιοι είναι τα θύματα και μετά να πάρουμε μια απόφαση που να βασίζεται σε μια καλή ε, λεπτομερή ανάλυση. Όχι, δεν έχω καμία διάθεση να πω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε τεχνολογίες, αυτό το σχέδιο κλπ. Αλλά εδώ πέρα είναι ένας οδοστρωτήρας που μας πρόχνει και μας σωθεί και ισοπεδώνει τα πάντα. Εδώ λοιπόν ε, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ηγετική θέση σε άλλα τεχνολογικά θέματα που πριν από τα 50, 60, 70 χρόνια θα μας δώσει ένα καρπό από ό,τι μας υπόσχονται εδώ με την πυρηνική σύνδεξη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ που ήρθατε κυρία και κύριοι Υπουργέ και μας είπατε τι μπορούμε να αναμένουμε μέχρι το τέλος του έτους. Μας είπατε ποιοι είναι οι σημαντικοί φάκελοι. Και βεβαίως ε, εγώ ενδιαφέρομαι κυρίως για την, ε, στρατη, για την πολιτική, τη βιομηχανική και για τη στρατηγική των α, ε, πρώτων υλών. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα κατευθύνεται τα πράγματα αυτά γιατί αυτά σχετίζονται κατά την άποψή μου πάρα πολύ στενά μεταξύ τους και για την πολιτική της έρευνας και της επιστήμης τι θα κάνετε εδώ πέρα γιατί νομίζω πως η έβρεση εναλλακτικών σε κάποιους σε κάποια πάρα πολύ σπάνια μέταλλα και πρώτες ύλες είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε υποκατάσταση και βεβαίως θα έχουμε και την ανακύκλωση όλων αυτών των ε, υλικών. Πρέπει να ενσωματωθούν όλα αυτά στην πολιτική. Κατόπιν ένα άλλο θέμα η ανάγκη ανταγωνισμού και η βιομηχανική πολιτική το οποίο είναι πάρα πολύ όπως είπε και ο κ. Ε, Λάγκε πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό σε ένα ευρύτατο πλαίσιο νομίζω πως ε, που και που γίνεται πρέπει να έρονται τα εμπόδια μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Δηλαδή η βιομηχανία σχετίζεται και με το εμπόριο και με την έρευνα και με την επιστήμη. Όλα αυτά πάνε μαζί γιατί για μένα ε, η ανταγωνιστικότητα σημαίνει μείωση και του ρυθμιστικού βάρους ε, και το πώς θα έχουμε ενιαίους κανόνες για την επιχειρηματική ζωή στην Ευρώπη. Γιατί εξακολουθούμε να έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα κανόνων. Ποτέ λοιπόν δεν ε, θα φτάσουμε στο επίπεδο που έχουν πύχει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η πολιτική μας. Ευχαριστώ κύριε Καρβάγιο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί, πρώτα-πρώτα, καλή τύχη. Και συγχαρητήρια για την Προεδρία σας, πάρα πολύ ρεαλιστικά. Ασκείτε τα κοντά σας, τώρα σας ευχαριστούμε που ήρθατε να μας παρουσιάσετε αυτές τις πρωτοβουλίες, συμφωνούμε και για την ψηφιακή να τη συμφωνούμε και για όλα όσα είπατε. Πρώτα πρώτα κύριε Λαριουέλ, έχω μία ερώτηση. Εσείς, από πλευρά πρακτικής, πώς βλέπετε να γίνεται αυτή η προοδευτική ένταξη, ε, συγχώνευση ας πούμε ESA και της κοινότητας. Ε, υπάρχει άλλη κουλτούρα, άλλη διάρθρωση, άλλα προγράμματα, άλλη χρηματοδότηση. Άρα πώς θα τα καταφέρουμε στην πράξη να κάνουμε ε, αυτό το οποίο θέλουμε και έτσι να έχουμε ενιαία διαχείριση. Τώρα για την χρηματοδότηση, κυρία Υπουργέ, μας είπατε για την Ίτερ μας είπατε για τον Γαλιλαίο και για το GMS έχουμε και το πρόγραμμα για την Αφρική πάρα πολύ χρήσιμο και συμφωνώ μαζί σας πέστε μας όμως πως θα μπορέσουμε όλα αυτά τα μεγάλα προγράμματα να τα καλύψουμε από χρηματοδοτικής Κύριε Υπουργέ τώρα, Πώς θα χρησιμοποιήσουμε ε, τους πόρους που υπάρχουν για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Όσον αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ε, ανάκαμψης, ήδη χρησιμοποιούμε ε, κάποιους πόρους, αυτά τα συγκεκριμένα ταμεία, ε, για αυτό το recovery plan. Όμως ε, για την Ήπεθρο έχουμε θέματα χαμηλής απορρόφησης, έχουμε συναρμοδιότητα πολλών τμήματων της Κομισιόν άρα να χρησιμοποιήσω όλο ένα περισσότερο ε, αυτά τα ταμεία την άψη της υπαίθρου, αυτούς τους πόρους για την προσβασιμότητα στην ε, πληροφορία πώς νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την καλύτερη αξιοποίηση Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημα απευθύνεται στην κυρία Υπουργό, την κυρία Ραουλιέλ. Σήμερα ψηφίσαμε τον προπολογισμό του 2011 και παρατήρησα με τρόμο πως υπάρχει πρόταση Κομισιών και Συμβουλίου να περιοριστεί, να περικοπεί το πρόγραμμα CIP για καινοτομία και έρευνα κατά δύο τρίτα. Ε, ελπίζω να μην γίνουν αυτές οι περικοπές. Ακριβώς σε σημερινές, ε, σημερινές συνθήκες πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το πρόγραμμα CRAFT για τις έρευνες ε, είναι για εμάς μεγάλη πρόκληση. Νομίζω θα μπορούσατε ίσως να αναλάβετε μια πρωτοβουλία για την πραγματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις μικρές Επιχειρήσει, Νομίζω πως ειδικά στην ε, Κομισιόν χρειάζονται εδώ πέρα νέες κατευθύνσεις. Δεύτερον, προς τον κύριο Υπουργό, σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία σας, για την ευρυζωνικότητα. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά στον τομέα του roaming. Πράγματι, έχετε δίκιο, ένα MB κοστίζει κατά κανόνα 2,6 ευρώ. Και στο, στη τιμή χοντρικής είναι 0,1 Send. Ε, δεν είναι αποδεκτό αυτό. Το συζητήσαμε σήμερα πως θα ήταν καλύτερο στο δίκτυο τέταρτης γενεάς να μην επιτρέψουμε ευθύς εξ αρχής χρεώσεις roaming, περιαγωγής. Να μην έχουμε λοιπόν τέτοιο ζήτημα καν να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και να πούμε LTE, το δίκτυο τέταρτης γενιάς, να έχει μία χρέωση εσωτερικής αγοράς και τέλος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργή, και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξή. Είναι δύο θέματα που νομίζω είναι πολύ σημαντικά. Μπορείτε να μου εξηγήσετε περισσότερο. Πρώτα πρώτα για τις ΜΜΕ. Στη σημερινή συγκυρία τη κρίση, ε, οι ΜΜΕ περνάνε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, ιδίω όσον αφορά το βιομηχανικό κλάδο. Και επίσης ε, μιλούμε τώρα για μια βιώσιμη ανάπτυξη και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιε αντιφάσει μεταξύ των κοινωνικών πολιτικών για ε, τις ε, ενισχύσεις της οικονομικές όσον αφορά την καινοτομία και κάποιες άλλες πιο συγκεκριμένες, πιο στοχευμένες ενισχύσεις όσον αφορά τις επενδύσεις των ΜΜΕ. Επίσης, πέστε μας εάν ε, προβλέπετε κάποια πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την δυσμενή κατάσταση και δυσμενές κλίμα που υπάρχει τώρα σαν φρακιά καινοτομία και ψηλόν. Τώρα για την ψηφιακή ατζέντα, κύριε Υπουργέ. Για το 2013 ε, θα πρέπει να έχουμε βριζονικές εφαρμογές για όλους Αυτό θα πρέπει να ισχύσει στην πράξη και μην μιλούμε μόνο για την ύπαθρο γιατί το 20% των Ευρωπαίων έχουν εισόδημα κάτω από το κατοφλή της φτώχειας και αυτοί θα πρέπει να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην ευρυζωνική ε, ψηφιακή ε, πραγματικότητα. Τι θα κάνετε τόσο ώστε να εξασφαλίσετε ότι σε όλο τον κόσμο θα προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ, κυρία Τόμψεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο υπουργού. Πολύ ενδιαφέροντα τόσο, μας είπαν. Πολύ σημαντικές αυτές οι προτεραιότητες. Και έτσι θα έχουμε την Ευρώπη της γνώσης. Τώρα όσον αφορά την διαστημική έρευνα, γενικά το διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πώς αλλάζει το κλίμα. Όσο θα ότι και εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε μια ομάδα δικού ενδιαφέροντο που ασχολείται με το διάστημα. Σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση τώρα, για πέστε μας. Τι γίνεται με τις επενδύσεις στην βιομηχανία. Γιατί η εμπειρία μας από τον Γαλιλαίο έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει κανείς ε, την βιομηχανία να κάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ακόμα και κάτι άλλο. Δεσμήμοι ε, γενικά για το επιχειρηματικό πνεύμα. Χρειάζεται περισσότερη ενθάρρυνση αυτών που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. το Φεβρουάριο του 2004 εκπώνησε ένα πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τότε όμως, και αφού υπευθύνει στα κράτη-μέλη, δεν γίνανε και πολλά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών, διότι οι όροι προποθέσει ε, συγκρότηση μια καινούργια επιχείρηση διαφέρει από χώρα σε χώρα. το Βέλγιο όσο αφορά την κοινωνική πολιτική είναι πρωτοπόρο. Χρειαζόμαστε επομένω τέτοια πρότυπα και να δούμε τι θα γίνει και με το δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί έτσι που συλλογίζονται τα πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε το, το ίδιο επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας στο μέλλον. Εσείς, τι προτίθεστε να κάνετε όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Κύριε Υπουργέ. Για πέστε μας για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Εγώ σαν ώρα με έχω ότι θα πρέπει να καλυφθεί όλη η Ευρώπη και χωρίς καλωδίωση. Δυστυχώς. Έχω μιλήσει στο Κόλμη με ένα επιστημονικό Ινστιτούτο ε, με κάποιους καθηγητές που είπαν ότι υπάρχουν δεσμενείς επιπτώσεις από τις ε, υπηρεσίες ε, wireless. Άρα εσείς όσον αφορά την παροχή των ευρωζωνικών υπηρεσιών χωρίς καλωδίωση wireless, πώς θα, τι θετικά θα για τις δεσμενείς επιπτώσεις. κυρία Φανμπρέντ, ευχαριστώ ορίζω και τους δύο υπουργού. Θα είμαι σύντομη γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Δύο ερωτήσεις στον κύριο Μπόρνε για το roaming δεδομένων το οποίο αναφέρατε. Ξέρω πως σας απασχολεί. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε και να είμαστε και αποτελεσματικοί. Και το ερώτημά μου σε εσά είναι τι θα α, προτιμήσετε γιατί βεβαίως αυτές τις τεράστιες διαφορές αγοράς σχετίζονται με τα κενά της αγοράς. Πρέπει λοιπόν να δουλέψει καλύτερα ο ανταγωνισμός ή πρέπει να ορίσουμε εμείς μέγιστες τιμές α, όπως έχουμε στο νερό και στον ηλεκτρισμό να ορίσουμε μέγιστες τιμές και γι' αυτό για το roaming δεδομένων. Και δεύτερο ερώτημα που σχετίζεται με το ερώτημα της κυρίας Τόμσεν. Οπωσδήποτε συμφωνείτε πως ε, είναι τόσο σημαντικές οι τηλεπικοινωνίες που είναι ένα είδος βασικού θα έλεγα δικαιώματος όπως το νερό, το ρεύμα και η στέγαση. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι' αυτό. Ευχαριστώ κυρία Τράουτμαν. Monsieur Président. Euh, voudrais Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στους ε, κυρίους υπουργούς ότι ε, αυτό είναι μια νέα πνοή αυτές οι πρωτοβουλίες ε, είναι το, το οξυγόνο για να μπορέσουμε να βγούμε από την ε, οικονομική κρίση με συγκεκριμένες δράσεις και μας μιλήσατε για την ε, ψηφιακή ατζέντα και τις άλλες και όταν μας μιλήσατε για το διάστημα, για τους δορυφόρους, για τα μέσα που θα αναπτυχθούν, για το φάσμα, για τις τηλεπικοινωνίες ότι υπάρχει εδώ πέρα μια λογική, ε, μια συνοχή αυτών μεταξύ τους που θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε. Για ε, να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το, χρονοδιάγραμμα όμως για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες. Ε, έχουν πλεονέκτημα έναντι των, ε, των ε, οπότε θα πρέπει και εμείς αυτό να εκμεταλλευτούμε όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου κλπ. Ε, συμφωνώ με όσο είπε ο κ. Ρούμπη και επαυξάνω όσον αφορά τις κοινωνικές ανισότητες αν ε, δεν προχωρήσουμε με οπτικές σύνες, με δορυφόρους, με, την, ε, με τις ευρωζωνικές υπηρεσίες θα μείνουμε πίσω. Να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο δυναμικά να προωθήσει τις ε, προτάσεις της για τους μη κυβερνικού οργανισμούς. Καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Θα πρέπει τα πράγματα να τα έχουμε καθαρίσει πριν αρχίσει για τον προπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για το Ταμείο Ανάπτυξης Πέθρου προηγουμένως. Δεν μπορούμε, εάν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, τι θέλουμε. Αν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεων. Γιατί το κλειδί της πολιτικής της επιτυχίας της είναι η καινοτομία, η πληροφορία, η βιομηχανία και η καινοτομία. Επομένως, να προσέξετε επίσης τα εξής. Πρώτον, η ουδετερότητα του δικτύου γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σχετικά με το άκτα τι γίνεται με τους ε, προμηθευτές αυτό θα πρέπει να το προσέξετε στις διαπραγματεύσεις και να προσέξετε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Τεχνολογίας όσον αφορά ε, τους ε, θύλακες και αν μπορείτε επομένως προσπαθήστε να με καλύψετε σήμερα. Ευχαριστώ, ακούσαμε όλα τα ερωτήματα. Θέλω να δώσω τώρα στους υπουργούς την ε, ερω... τη δυνατότητα να απαντήσουν. Θα ελπίζω να μας δώσουν λίγο χρόνο και οι αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε γρήγοροι. Κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές ήταν οι ερωτήσεις για πολλά θέματα και καταλαβαίνω πως νιώθουν απογοητευμένοι μερικοί. Μια που έχουμε αυτή την κατανομή ε, των αρμοδιοτήτων στο βελγικό κράτος και είπατε ότι Άλλος σχολεί με καινοτομία, άλλο με, με την ανταγωνιστικότητα, αλλά θα πρέπει να σας καλύψουν για το ίδιο θέμα. Αλλά μη φοβάστε. Θα, θα, θα, θα σας ικανοποιήσουμε τα ερωτήματα. Σήμερα είπαμε να συζητήσουμε το διάστημα. Και είπαμε από την άλλη μεριά ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι πιο ανταγωνιστικές η ΜΜΕ. Βεβαίως είναι δικό μου χαρτοφυλάκιο και με ενδιαφέρει. Να σας πω δύο λόγια. Με δεδομένη την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών Υπουργείων. Κύριε Λάμπερτ, εγώ όχι, δεν θέλω μαζί με τα ξερά να κάνουν και τα χλωρά. Γιατί ο αυτό το ίτερ, έχουμε πολλές απόψεις του θέματος έχουμε το GMS, έχουμε το Galileo, έχουμε λοιπόν τρία θέματα τα οποία απασχολούν την ε, Βελική Προεδρία. Είναι θέμα δημοσιονομικό όπου έχουμε πρόβλημα. Και για τα τρία αυτά προγράμματα που μας έχουμε ενδιαφέρον.